Καλησπέρα σας συνάδελφοι. Παρακαλώ καθίστε για να μπορέσουμε να ξεκινήσουμε. Όπως ξέρετε, έχουμε μια κοινή συνεδρίαση των Επιτροπών Οικονομικών και Νομισματικών Υποθέσεων και Προϋπολογισμών βάσει του άρθρου 55. Καταρχά να εγκρίνουμε την ημερήσια διάταξη, δεν υπάρχουν παρατηρήσεις, σα ευχαριστώ. Δεν έχω ανακοινώσει να κάνω, οπότε μπορούμε απευθεία να περάσουμε στο σημείο 3. Δημόσια ακρόαση για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων. Ένα θέμα ιδιαίτερα επίκαιρο στην όλη διαδικασία ετοιμασίας και σύνταξης της έκθεσης σε βάση της κλασικής νομοθετικής διαδικασίας και βάσει των όσων υπέβαλε ως προτάσεις η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να υπάρξει ανάκαμψη των επενδύσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είχαμε μια πολύ επικοδομητική συνάντηση διαλόγου και ρωταπαντήσεων με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή την περασμένη εβδομάδα. Τις επόμενες ημέρες ο εισηγητή θα περατώσει τη σύνταξη τη έκθεσης, οπότε είναι ευπρόσδεκτη αυτή η ευκαιρία να συζητήσουμε κάποια ζωτικά σημεία του προγράμματος Juncker. με κάποιους εξέχοντες εμπειρογνώμονες. Έχουμε διαιρέσει την ακρόαση σε δύο τμήματα στην, ε, στο πρώτο μέρος της ε, ακρόασης θα, προεδρεύσει, θα προεδρεύσω εγώ ίδιος, στο δεύτερο μέρος ο κύριος Αρτουή. Στο πρώτο μέρος της ακρόασης θα επικεντρωθούμε στο μακροοικονομικό αντίκτυπο. Θεωρούμε ότι θα υπάρξει, δεν είναι κάτι δεδομένο βέβαια το τι ακριβώς θα συμβεί με το πρόγραμμα, και το σημαντικό θέμα της διακυβέρνησης του ταμείου αυτού, του νέου ταμείου, το θέμα της επιλογής των έργων και εξίσου σημαντικό και τελευταίο την απαραίτητη προϋπόθεση που όλοι επιζητούμε είναι η σωρευτικότητα, η προστατικότητα της χρηματοδότησης του Ταμείου. Πώς θα την εξασφαλίσουμε. Αυτό έχει να κάνει βεβαίως και με τι διατάξει του κανονισμού, με το σύστημα διακυβέρνησης που θα προβλεφθεί για το Ταμείο, τα υπόλοιπα, έργα, το, τα υπόλοιπα όργανα μάλλον, τα συμβουλευτικά και τα κριτήρια που θα ορίσουμε σχετικά. Όλα αυτά θα πρέπει να καταρτιστούν στη συμφωνία που θα ιδρύει το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στατικών Επενδύσεων. Να ξεκινήσουμε δίνοντας το λόγο στον πρώτο ομιλητή του πρώτου πάνελ, 10 λεπτά στον καθένα. Μετά θα δώσουμε το λόγο στους συζητητές και μετά και πάλι στους προσκεκλημένους ομιλητές μας για τις απαντήσεις τους. Και μετά στους υπόλοιπους ε, αγορητές της ε, κάθε επιτροπής. Πριν ξεκινήσω, να δώσω το λόγο στο Ζαν. Θες κάτι να προσθέσεις. Ευχαριστώ. Ναι, δεν χρειάζεται να προσθέσω τίποτα. Καλύτερα να περάσουμε αμέσως στην ακρόαση. Καλώς, αρχίζουμε με τον πρώτο μιλητή τότε. Είμαστε πολύ περήφανοι που έχουμε μαζί μας τον Φίλιπ Μάιστατ, που είναι ως πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Έχεις το λόγο, Φιλίπ. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, δύο προκαταρκτικές ε, παρατηρήσεις. Πρώτο, είμαι πεπισμένος ότι το σχέδιο επενδύσεων Juncker θα καταδείξει και είναι μια πρώτη ετάπ, ένα πρώτο στάδιο για την ευαισθητοποίηση της αναγκαιότητας να επενδυθούν περισσότερα σε υποδομές και στις βιομηχανίες της αύριο. Μπορεί βέβαια κανείς να επικρίνει το σχέδιο και μάλιστα και εγώ έχω κάποιες κριτικές παρατηρήσεις για το σχέδιο επενδύσεων. Ωστόσο, το κάνω μέσα σε ένα επικοδομητικό πνεύμα, γιατί μου φαίνεται πραγματικά επιτακτικό να επιτύχει το σχέδιο μέσα στο παρόν πολιτικό κλίμα όπου καμιά φορά αμφισβητείται η πολιτική και η στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι σημαντικό λοιπόν η Ευρωπαϊκή Ένωση να καταδείξει ότι ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα μπορεί να έχει θετική επίπτωση, βραχυπρόθεσμα στην ζήτηση, διότι οι επενδύσεις θα δώσουν δουλειά στις επιχειρήσεις που θα φτιάξουν μετά τις υποδομές που θα κατασκευάσουν τους απαραίτητους εξοπλισμούς, θα προωθήσουν προγράμματα έρευνας και από την άλλη μεριά πιο μακροπρόθεσμα από την πλευρά της προσφοράς και επομένως και της ανάπτυξης. Άρα πρώτο είναι απαραίτητο να γίνει κάθε τι το δυνατό για να επιτύχει το σχέδιο Juncker. Δεύτερη προκατακτική παρατήρηση. Γνωρίζετε ότι το σχέδιο Juncker βασίζεται σε τρεις πυλώνες. Υπάρχει ο πυλώνας για τον οποίο θα μιλήσουμε σήμερα, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων. Μην λησμονούμε όμως ότι υπάρχει και ένας δεύτερος πυλώνας που είναι η κοινή πλατφόρμα τεχνικής βοήθειας για τα διάφορα έργα και τρίτος πυλώνας που είναι η προώθηση της ενιαίας αγοράς σε ορισμένους τομείς κλειδιά όπως ενέργεια, μεταφορές και ψηφιακή τεχνολογία. Ο δε Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Κατάινεν επαναλαμβάνει διαρκώς ότι στα μάτια του ο τρίτο πυλώνας είναι μάλιστα πιο σημαντικός και σίγουρα έχει δίκιο. Όμως πρέπει κανείς να ελπίσει ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα προχωρήσει πολύ σύντομα σε κατάθεση προτάσεων για τον τρίτο πυλώνα. Τώρα, με αυτές τις δύο προκατακτικέ παρατηρήσεις θα ήθελα να έρθω, σύντομα βέβαια, γιατί μα ζητήσατε να περιοριστούμε σε 10 λεπτά, να έρθω λοιπόν βέβαια με τρόπο συνοπτικό στο θέμα. Βεβαίως μπορώ να πω σε περισσότερες λεπτομέρειες όταν θα τεθούν ερωτήσεις. Το πρώτο λοιπόν είναι βέβαια το θέμα της προσθετικότητας. Εδώ υπάρχουν δύο πτυχές. Για να υπάρξει βέβαια θετική επίπτωση στην οικονομία πρέπει να είναι πρόσθετες συμπληρωματικές επενδύσεις. Δηλαδή επενδύσεις που δεν θα γίνουν χωρίς το πρόγραμμα Juncker. Εδώ υπάρχουν δύο πτυχές όπως είπα. Αφενός τα 16 δισεκατομμύρια που θα δεσμεύσει η Ευρωπαϊκή Ένωση για το Ταμείο Εγγύσεων να προβλεφθούν τουλάχιστον εν μέρη στον κοινοτικό προϋπολογισμό στην διευκόλυνση συνδέοντα στην Ευρώπη και στον ορίζοντα 2020 για την έρευνα. Τα περίφημα άρθρα 18 και 19 του σχεδίου κανονισμού. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λέει ότι οι πιστώσεις που θα μεταφερθούν έτσι θα έχουν σημαντικότερη επίπτωση εάν περάσουν μέσα από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στατικών Επενδύσεων. Ίσως, αλλά αυτό χρειάζεται επαλήθευση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λέει ότι θα προχωρήσει την επαλήθευση. Δεν έχει εξηγήσει ακόμα πώς θα κάνει την επαλήθευση αυτή. Ίσως υπάρχουν κάποιες δυσκολίες μεθοδολογικού χαρακτήρα για να διασφαλίσει ότι όντως θα υπάρξει σημαντικότερο αποτέλεσμα. Για τις πιστώσεις εκείνες που αρχικά επαναλαμβάνω, προβλέπονταν ως στήριξη των ε, δημοσιονομικών εργαλείων. Το δεύτερο, η δεύτερη πτυχή της υποστατικότητας είναι ότι πρέπει να διασφαλιστεί ότι η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων δεν πρόκειται να χρηματοδοτήσει μέσω του ΕΦΣΥ τις επενδύσεις που ούτως ή άλλως θα ε, χρηματοδοτούνταν από τις συνήθεις εργασίες της. Υπάρχει τώρα και το στοιχείο του κινδύνου. Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων έχει αλλάξει πολύ αναλαμβάνει μεγαλύτερο κίνδυνο σήμερα από ότι εδώ και 20 χρόνια αλλά έχει και λόγους να το πράξει αυτό. Θέλει να διατηρήσει την βαθμολόγησή της τριπλού α. Λένε πολλοί ότι έχει ακόμα μεγαλύτερη σημασία από το τριπλό α. Θα σας εξηγήσω όμως γιατί είναι σημαντικό να διατηρήσει την βαθμολόγηση αυτή. Ένα επιχείρημα είναι ότι η βασική κατηγορία αγοραστών των ομολόγων της ΕΤΕ είναι οι κεντρικέ τράπεζε σε όλο τον κόσμο. Οι μεγαλύτεροι δηλαδή αγοραστέ ομολόγων. Αν πέσει από το τριπλό α στο 2α η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων θα σταματήσουν οι κεντρικές τράπεζες από ανταχού του κόσμου να αγοράζουν τα ομολογά τη. Είναι λοιπόν φυσιολογικό η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων να προσέχει πάρα του κινδύνου που αναλαμβάνει. Ακριβώ όμω το σχέδιο Juncker τη δίνει την ευκαιρία να, να αναλάβει μάλλον περισσότερου κινδύνου. Για μένα είναι σαφές ότι χρειάζεται μια δέσμευση της ΕΤΕ ότι θα χρησιμοποιήσει το Ευρωπαϊκό ε, Ταμείο Στατικών Επενδύσεων για να, για επενδύσει σε πιο σε, σε, σε έργα με μεγαλύτερο κίνδυνο από ότι αυτά που συνήθως χρηματοδοτεί. Δεύτερον, αυτό το περίφημο, αυτή η περίφημη μόχλευση που φαίνεται σημαντική, φιλόδοξη. Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων ήδη έχει επιτύχει μια σημαντική μόχλευση στο παρελθόν. Με διαφορετικούς όρους όμως. Για παράδειγμα, από τα πρώτα προγράμματα ήταν η Risk Sharing Facility για την έρευνα, που μετά έγινε πρόγραμμα μέσα στην ε, δημοσιονομική προοπτική, 3 δισεκατομμύρια εγγυήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης που επιτρέπει στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων να δανείσει 18 δισεκατομμύρια, επομένως 1 προς 6 και αυτά τα 18 δισεκατομμύρια μπορούν τελικά να επιτρέψουν μια συνολική χρηματοδότηση 48 δισεκατομμυρίων. Επομένω εδώ η μόχλευση είναι πιο σημαντική. Αλλά βλέπετε ποιε είναι οι αναλογίε. Είναι αρκετά διαφορετικέ από αυτέ που προβλέπονται στο σχέδιο Juncker. Οπωσδήποτε υπάρχει ένα πράγμα που μου φαίνεται βέβαιο. Ότι δεν θα καταφέρουμε να προσελκύσουμε ιδιώτε επενδυτέ τουλάχιστον με την προβλεπόμενη αναλογία. Δηλαδή για τα 4 πέμπτα τέσσερα πέμπτα να προέρθουν από ιδιωτικέ επενδύσει. Δεν θα καταφέρετε λοιπόν να προσελκύσετε του ιδιώτε επενδυτέ εάν του μεταχειριστείτε λιγότερο καλά από ότι την ε, Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Έτσι λοιπόν, μέσα στο σχέδιο κανονισμού που σα έχει υποβληθεί, η, εγγύηση, η ευρωπαϊκή εγγύηση δίνεται μόνο στην ΕΤΕ. Δεν λαμβάνει υπόψη του ε, ιδιώτε επενδυτέ. Ο μόνο τρόπο για να γίνει ελκυστικό το πρόγραμμα αυτό για τον ιδιωτικό κλάδο είναι να ζητήσετε ώστε η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων γενικά να λαμβάνει μια θέση junior, δηλαδή να παρεμβαίνει με εργαλεία χαμηλότερης κατηγορίας από τους ιδιώτες επενδυτές. Γιατί αλλιώς θα πούν, μα κοιτάξτε εσείς ε, εγγυάστε την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, αλλά δεν εγγυάστε τις ιδιωτικές επενδύσεις. Νομίζω ότι έχουν την πρόθεση αυτή, αλλά νομίζω ότι δεν είναι και άχρηστο να δηλωθεί ρητά η πρόθεση αυτή, είτε στον κανονισμό, είτε στη συμφωνία μεταξύ ε, Ευρωπαϊκής Επιτροπής και Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Δεύτερο, η διακυβέρνηση, governance. Θα προχωρήσω με ταχύτητα βέβαια, γνωρίζετε όμως και το περιεχόμενο των προτάσεων. Υπάρχει ε, η Διευθύνουσα Επιτροπή Διαχείρισης και τα όργανα της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Για το νομικό θέμα δεν μπορεί να τροποποιήσει κανείς τις διαδικασίες λήψους αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων όπως αυτές καθορίζονται από το πρωτόκολλο που έχει προσαρτηθεί στις συνθήκες. Πρέπει να παραμείνει μέσα στα πλαίσια των συνθήκων. Νομίζω επίσης ότι πρέπει να γίνει μια διάκριση μεταξύ του ρόλου της Διευθύνουσας Επιτροπής που θα δίνει κάποιες γενικές κατευθύνσεις της πολιτικής επενδύσεων για το προφίλ των κινδύνων του συνολικού χαρτοφυλακίου. Αυτός θα είναι ο ρόλος αυτής της Piloting Committee και αυτό νομίζω, εκεί νομίζω ότι πρέπει να ασκηθεί ο κοινοβουλευτικός έλεγχος από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και μετά έρχεται η επιλογή των μεμονωμένων έργων. Αυτή η επιλογή των μεμονωμένων έργων θα πρέπει να παραμείνει, πιστεύω, υπόθεση της ίδιας της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων που είναι πολύ καλύτερα εξοπλισμένη για την επιλογή των έργων που θα είναι πλέον βιώσιμα και πλέον στέρεα. Και ποιος είναι τώρα ο ρόλος της Επιτροπής Επενδύσεων. Εγώ θα ήθελα μάλιστα να δω πώς εξελίσσεται το κείμενο του σχεδίου κανονισμού. Ήδη έχει αλλάξει πολύ. Νομίζω πάντως ότι ο ρόλος της Επιτροπής Επενδύσεων που θα αποτελείται όπως γνωρίζετε από έξι ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες δεν θα είναι να επιλέξει τα ίδια τα έργα διότι πώς και να το πράξει και οι πιο μεγάλοι ειδικοί και αν είναι μόνο έξι δεν μπορούν να το κάνουν αυτό. Ο ρόλος αυτής της Επιτροπής Επενδύσεων θα πρέπει να είναι να επαληθεύει εάν τα έργα που επιλέγει η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων ανταποκρίνονται στις προϋποθέσεις του άρθρου 5 του σχεδίου κανονισμού και στους προσανατολισμούς, τις πολιτικές, το προφίλ ρίσκου που καθορίζει η ε, Διευθύνουσα Επιτροπή. Εφόσον έχει δικαίωμα σε ευρωπαϊκές εγγύησεις, θα πρέπει να τα αποκρίνεται στους όρους αυτούς. Τέταρτο θέμα, η εγγύηση. Ακόμα συζητείται το θέμα αυτό. Κατανοώ βέβαια την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που θέλει να αποζημιώνεται για, τον, για το ρίσκο που αναλαμβάνει, επομένως ο κοινοτικός προπολογισμό και θα θέλει μια ανταμοιβή όσο γίνεται υψηλότερη από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων πρέπει λοιπόν πρέπει να παραμείνει κανείς λογικός μέσα σε αυτό το πλαίσιο. Πέμπτο ερώτημα. Εξετάζοντας την λίστα των επενδύσεων που ενδέχεται να χρηματοδοτηθούν από το ΕΦΣΙ, από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στατικών Επενδύσεων, είναι σαφές ότι ο ένας αριθμός από τα έργα αυτά ποτέ δεν θα προσελκύσουν τέσσερα πέμπτα χρηματοδοτήσεως από τον ιδιωτικό τομέα. Είναι σαφές για μένα αυτό, διότι πρόκειται για έργα τα οποία βεβαίως είναι σημαντικά και ενδιαφέροντα, έχουν μια απόδοση κοινωνική ή και οικονομική καμιά φορά σημαντική, αλλά η οικονομική απόδοση πολύ ασθενή ή πολύ αβέβαια ή πολύ μακροπρόθεσμη. Δεν πρόκειται λοιπόν να προσελκύσουν τα ιδιωτικά κεφάλαια. Αρκετά σημαντικό αριθμό λοιπόν των σχεδίων αυτών έχει περισσότερη, θα χρειαστεί περισσότερη δημόσια στήριξη. Εδώ σας επισημαίνω το εξή, ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το γνωρίζει αυτό και το γράφει μάλιστα και ρητά σε άλλο έγγραφο που δημοσίευσε για την Ένωση των Κεφαλαίων. Ότι ορισμένα έργα θα χρειαστούν περισσότερη δημόσια στήριξη εκ της φύσεώς τους. Το αναγνωρίζει αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και αυτό που κάνει είναι ότι προσφέρει διευκρινήσεις για την εφαρμογή των κανόνων του Συμφώνου Σταθερότητας και πιο συγκεκριμένα για αυτό που ε, ονομάζει ρήτρα επενδύσεων μέσα στα πλαίσια του Συμφώνου Σταθερότητας. Δηλαδή τη δυνατότητα μιας προσωρινής παρέκκλησης από την τροχιά της προσαρμογής για τους μεσοπρόθεσμους στόχους σταθερότητας, γνωρίζετε ότι είναι υποχρεωτικό να τηρηθεί αυτή η τροχιά, όταν θα εποφελείται κανείς από τη ρήτρα αυτή θα μπορεί να έχει μια προσωρινή παρέκκληση. Προσθέτει όμως το ίδιο έγγραφο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι πρέπει να πληρούνται ορισμένες προϋποθέσεις για να επωφεληθεί κανείς από τη ρήτρα αυτή. Και μεταξύ των προϋποθέσεων αυτών είναι και ότι το ενδιαφερόμενο κράτος δεν μπορεί να έχει έλλειμμα μεγαλύτερο του 3% του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος. Υπό τις παρούσες συνθήκες είναι σαφές ότι ένας συγκεκριμένος αριθμός χωρών μελών, και γνωρίζετε για ποιες μιλώ, και η χώρα του Προέδρου μας αποκλείονται αυτομάτως από το ευεργέτημα της ρήτρας αυτής. Σας επισημαίνω λοιπόν αυτή την πτυχή. Προσωπική μου άποψη είναι ότι εφόσον πρόκειται για μια επένδυση που έχει αναλυθεί σε βάθος από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων, που έχει εγκριθεί από τα όργανα της Ευρωπαϊκής Τραπέζης Επενδύσεων και χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων, η ενδεχόμενη δημόσια συγχρηματοδότηση θα πρέπει να μπορεί να υποφεληθεί από την ρήτρα επενδύσεων χωρίς παραπέρα ιστορίες. Το άλλο διακόπτει ο πρόεδρος Γκουαρτιέρη. Σας παρακαλώ να ολοκληρώσετε πιο σύντομα. Η συνεργασία με τις ε, δημόσιες τράπεζες, το ιδεώδες θα ήταν να συμβάλλουν στο ΕΦΣΥ, αλλά για διαφόρους λόγους νομίζω δεν θα το πράξουν. Μπορούν ωστόσο να, να συμβάλλουν σε ένα ταμείο που θα συμβάλλει με τη σειρά του στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Στατικών Επενδύσεων. Και τελειώνοντας, τελευταίο ερώτημα, το έβδομο, το θέμα του κινδύνου να υπάρξει υπερβολική συγκέντρωση των επενδύσεων εννοείται σε ορισμένες χώρες μέλη. Διότι αφενός υπάρχει μια φυσική τάση της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων να αντιμετωπίζει πρώτα-πρώτα σχέδια όπου θα συγκεντρωθεί ένα σημαντικό όγκο των δυνατών συντομότερα. Δεύτερο, το γεγονό ότι οι, οι ιδιώτες επενδυτές μάλλον θα τείνουν να επενδύσουν περισσότερο σε ορισμένε χώρε. Τρίτο, οι κανόνε του ε, Συμφώνου σταθερότητα. Τέταρτο, το ότι οι κεντρικέ τράπεζε είναι ισχυρότερε σε ορισμένες χώρες μέλη από άλλε. Άρα υπάρχει κίνδυνο μια υπερβολικά μεγάλη συγκέντρωση των επενδύσεων σε ορισμένε χώρε μέλη. Σωστά λέει το σχέδιο Juncker, δεν υπάρχει εκ των προτέρων κατανομή γεωγραφική ή άλλη, αλλά νομίζω ότι πρέπει κανείς να λαμβάνει υπόψη και αυτό το στοιχείο της κατανομής των επενδύσεων του ΕΦΣΥ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Μάιστατ για... για την παρουσίασή σας. Τα σημεία που τονίσατε ήταν όντως ζωτικής σημασίας. Και τώρα ο λόγος στο Hans Bruins, εκτελεστικό διευθυντή στον οργανισμό τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, που μου δίνετε την ευκαιρία να συνεισφέρω σε, αυτό, σε αυτή την τόσο σημαντική ακρόαση και συζήτηση για το ΕΦΣΥ. Θα ήθελα στην παρουσίασή μου να τονίσω την ανάγκη χρηματοδότησης της μετάβασης σε μια πράσινη οικονομία που προ στιγμήν μπορούμε να στηρίξουμε μόνο με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Όλα αυτά σχετίζονται και με την πρόταση κανονισμού, όπου τα κριτήρια για την ανάπτυξη απαιτούν την έρευνα, την καινοτομία, τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, την ενεργειακή αποδοτικότητα και τις υποδομές για περιβαλλοντικούς σκοπού και περιβαλλοντικούς πόρους. Επόμενη διαφάνεια. Αυτά που θα πω θα βασιστούν στην πενταετή καταγραφή στοιχείων που έχουμε κάνει για το περιβάλλον, μια αποβολή εκθέσεων που θα αρχίσει επισήμω αύριο στι Βρυξέλλε, αλλά τα πορίσματά τη έχουν να κάνουν με τι προτεραιότητε των επενδύσεων που θα προβλέψουμε για να μην ε, διασπαθήσουμε τους ισχνούς δημοσιονομικούς, κρατικούς και ιδιωτικού πόρους. Οι περιβαλλοντικές και κλιματικές πολιτικές έχουν δώσει σημαντικά ωφέλη για το περιβάλλον, αλλά και για την οικονομία και την υγεία των πολιτών και την ευμερία τους. Το δεύτερο βασικό πόρισμα είναι ότι η Ευρώπη αντιμετωπίζει, όπως και οι περισσότερες χώρες του πλανήτη, σοβαρές προκλήσεις προβλήματα σε ό,τι αφορά το σύστημα παραγωγής και κατανάλωσης που δεν είναι πλέον βιώσιμα στη μορφή τη σημερινή. Αλλάζουν και μεταβάλλονται ταχαίως στο σημερινό πλαίσιο. Εάν φανταστούμε ότι η παγκόσμια παραγωγή θα τριπλασιαστεί ως το 2050, τότε προφανώς οι σημερινοί πόροι και η χρήση της ενέργειας δεν μπορεί να, συνεχιστούν, να συνεχιστούν ως, ε, όπως τα γνωρίζαμε. Δεν είναι βιώσιμη αυτή η οδός για την περιβαλλοντική ανάπτυξη. Εάν θέλουμε να φτάσουμε τους στόχους του 2050 όπως έχουν οριστεί από τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και στο 7ο ε, πρόγραμμα δράση για το περιβάλλον αλλά και στο πακέτο για την ενέργεια και το κλίμα, στην πολιτική των μεταφορών και σε άλλους τομείς πολιτικής όπως την ε, οικονομία που θα είναι απαλλαγμένη από τον άνθρακα, την κυκλική οικονομία και το ισχυρό ε, εθνικό κεφάλαιο, θα πρέπει να αναζητήσουμε την οικονομική ευημερία αλλού. Δηλαδή, να περάσουμε σε αλλαγέ και μεταβάσει. Αυτό είναι ένα δυσχερέ εγχείρημα. Πιστεύουμε όμω ότι θα έχουμε έτσι τεράστιε ευκαιρίε για την οικονομία τη Ευρώπη και την απασχόληση και θα μπορέσει να φτάσει στην πρωτοπορία τη επιστήμη και τη καινοτομία η Ευρώπη. Επόμενη διαφάνεια. Αυτή η γραφική παράσταση είναι πολύ απλή και σαφής. Οι δύο χαμηλότερες γραμμές είναι το σύνολο του ΑΕΠ τη Ευρωπαϊκή Ένωση, η χαμηλότερη γραμμή είναι η εξέλιξη της απασχόλησης στην Ευρώπη. Από τη στιγμή που ξεκίνησε η κρίση το 2008, οι δύο ε, με πάνω γραμμές είναι η προστιθέμενη αξία στα περιβαλλοντικά αγαθά και ε, τις υπηρεσίες, τον σχετικό κλάδο και η γαλάζια γραμμή είναι οικολογικέ υπηρεσίε και αγαθά. Αυτά από τότε που ξεκίνησε η ύφεση στην Ευρώπη. Οπότε ο άμεσο συσχετισμό με τι φιλοδοξίε μα να αξιοποιήσουμε το ΕΦΣΙ για να υπερβούμε την οικονομική κρίση με μακροπρόθεσμη ενδυνάμωση τη Ευρώπη φαίνεται ξεκάθαρα από τη γραφική παράσταση. Φαίνεται την δρόμο έχουμε ακολουθήσει από το 2008. Επόμενη διαφάνεια. Εάν δούμε το μέλλον και τις λεπτομέρειες εδώ δεν πρέπει να τις ε, κοιτάξουμε ε, με επιμονή, η ουσία είναι ότι οι πόροι που θεωρήθηκαν κρίσιμοι, ε, κρίσιμες αξίες από την Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι ευρωπαϊκοί για το μέλλον. Οι κόκκινοι έρχονται από την Κίνα, οι υπόλοιποι από τη Βραζιλία, από την ε, Δημοκρατία του Κονγκό, τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό και άλλα σημεία στον πλανήτη. Όλα αυτά ε, συνάδουν με την πρόσφατη έκθεση του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ που λέει ότι τέσσερα Τέσσερι από του δέκα μεγαλύτερου κινδύνου για την οικονομία και τι επιχειρήσει έχουν να κάνουν με το κλίμα και το περιβάλλον. Όχι μακροπρόθεσμα μόνον, αλλά μέσα στην επόμενη δεκαετία. Οπότε το να επενδύσουμε σε ένα μέλλον που αυτού του κινδύνου του αναχαιτίζει, του καλύπτει, είναι κάτι που συμφωνεί με τι προτεραιότητε τη κυκλικής οικονομία και τη χαμηλή κατανάλωση άνθρακα. Θα ήταν μια ευθύ επιλογή και από την ε, σκοπιά του κινδύνου. Επόμενη διαφάνεια, ο σχετισμό με την χρηματοδότηση αυτή τη μετάβαση. Πρέπει να βρούμε δημοσιονομικούς πόρους είναι καθοριστική σημασία σε αυτό για την επίτευξη της οικονομίας που θα είναι απαλλαγμένη από τον άνθρακα και θα σέβεται την χρήση των πόρων. Αυτό έχει τονιστεί και από τον προηγούμενο ομιλητή. Οι εκτιμόμενες ανάγκες για ανάπτυξη προς την πράσινη οικονομία είναι τεράστιες. Η επικείμενη έκθεση των ευρωπαϊκών οργάνων μιλούν για δύο-τρει στον τομέα τη ενέργεια τα ερχόμενα 20 χρόνια και ο δικό χάρτη τη Ευρώπη για την οικονομία χαμηλή κατανάλωση άνθρακα μιλά για 217, 270 μάλλον δι τον χρόνο τα επόμενα 40 χρόνια. Είναι προφανέ ότι η δημόσια χρηματοδότηση θα, θα καθοριστικό ρόλο για την αναχέτηση των κινδύνων που αντιμετωπίζουν οι ιδιωτικοί επενδυτέ και για να ε, ενδυναμώσει την καινοτομία. Εδώ το Ευρωπαϊκό Στρατηγικό Ταμείο μπορεί να διαδραματίσει ένα σοβαρό ρόλο. Τα δημόσια κονδύλια από την έρευνα που έχει γίνει έχουν δώσει τι δυνατότητε να υπάρξει ρηξικέλευτη καινοτομία είτε στην φαρμακοβιομηχανία, είτε στην πληροφορική, είτε στην νανοτεχνολογία και σε όλε τι μορφέ τεχνολογία και με περιβαλλοντικέ ε, ανακαλύψει σε ό,τι αφορά τον κλάδο αυτό τη καινοτομία. Το θέμα είναι αν αυτή η πρόσθετη χρηματοδότηση μπορεί να αξιοποιηθεί για να φτάσει στην πορεία αναζήτηση των λύσεων εχμής ε, στην πράσινη τεχνολογία Ευρώπη. Η Ευρώπη ε, ε, έχει ένα μικρό μέρο του παγκόσμιου πληθυσμού προ ε, του ρυθμού ανάπτυξη. Μπορεί όμω η Ευρώπη να μετατραπεί σε Silicon Valley ε, ω προ τι ε, πράσινε τεχνολογίε με στήριξη των δημόσιων κονδυλίων και τα σχετικά κίνητρα. Επόμενη διαφάνεια. Η σταθερότητα και τα κίνητρα για τις πράσινες επενδύσεις είναι προφανώς ε, ουσιώδους σημασίας. τα πολιτικά πλαίσια καθορίζονται με τρόπο ώστε να συσχετίζουν τους στόχους που έχουμε σήμερα στην πολιτική και τις παρεμβάσεις που απαιτούνται. Το ΕΦΣΥ είναι μια τέτοια μεγάλη πολιτική παρέμβαση. Εάν θέλουμε μακροπρόθεσμα να έχουμε αποτέλεσμα και να υπάρξει σταθερότητα στον τομέα των ανεώσιμων λόγου χάρη, στην κυκλικότητα της οικονομίας, που είναι ε, επί της ουσίας ε, η χρήση των πόρων, υψηλή χρήση των πόρων και σχετική παραγωγικότητα, θα πρέπει όλα αυτά να τα δούμε από τη σκοπιά του 2020 και του 2050. Τότε αποκτούν την ιδιαίτερη σημασία τους. Ένα πρόσθετο στοιχείο είναι η σχέση με τις μετατοπίσεις της φορολόγησης. Η περιβαλλοντική φορολόγηση και σχετικές μεταρρυθμίσεις που έχουν να κάνουν με την χρήση των πόρων, την ρήπανση, αλλά και τις δημογραφικές εξελίξεις για τα φορολογικά συστήματα, είναι ένα ουσιαστικό στοιχείο. Ε, η σταδιακή εξάλληψη των επιζήμιων για το περιβάλλον επιδοτήσεων, καθώς και τα πρόσθετα κίνητρα χρηματοδότησης, ή η χρηση των ορυκτών καυσίμων, οι μηχανισμοί κινήτρων και οι μηχανισμοί επιδοτήσεων είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Έτσι, οι ευρωπαϊκοί περιβαλλοντικοί φορείς συστήνουν τα αυστηρά κριτήρια επιλογής για τις μελλοντικές επενδύσεις στην πράσινη οικονομία, βασιζόμενοι σε τέσσερα βασικά στοιχεία. Ένα είναι το κατά πόσον μπορούμε όντω να συμβάλλουμε στην απαλλαγή τη οικονομία από τον άνθρακα. Δεύτερον, κατά πόσον μπορούν να συμβάλλουν στην κυκλικότητα της οικονομία και άρα και στι ε, θέσει εργασίας για το μέλλον. Τρίτον, κατά πόσον προστατεύονται οι πράσινες υπηρεσίες, το οικολογικό κεφάλαιο και η κατάσταση του περιβάλλοντος σε πλανητικό επίπεδο με την ε, χαμηλή κατανάλωση ενέργειας. Και τέταρτον, κατά πόσον συμβάλλουν στην ανθρώπινη υγεία και ευημερία. Να περάσω τώρα στα αναμενόμενα ωφέλη στην επόμενη διαφάνεια. Τα αναμενόμενα ωφέλη από τις επενδύσεις στην πράσινη οικονομία και αυτό βασίζεται στα δικά μας μεν πορίσματα αλλά και στην διεξοδική έρευνα που έχει γίνει από, μεγάλους, από μεγάλα διεθνή ιδρύματα όπως ο ΣΑ και η Παγκόσμια Τράπεζα όλα αυτά δείχνουν ότι η απασχόληση κατά την οικονομική κρίση από το 2008 ως σήμερα επέτρεψαν την ανάπτυξη του, πράσινου τομέα από το 2,8 σε 4,1 εκατομμύρια θέσει εργασία. Αυτό είναι μια τεράστια εξέλιξη. Στην κοινοτομία από το 2008 έχουμε διάυξηση στι ε, τάσει τη Ευρώπη σε αυτόν τον τομέα. Ο τομέα έχει γίνει πιο ανταγωνιστικό από ό,τι στο παρελθόν, χάρη, μάλλον κατά τη διάρκεια τη περίοδου τη κρίση. Ε, η παραγωγικότητα ω προ τις των πόρων βελτιώθηκε η χρήση των πόρων ε, και η έλλειψή του είναι κάτι που θα απασχολήσει μια περισσότερη στην Ευρώπη. Πρέπει να καθορίσουμε μια μελλοντική στρατηγική. Εδώ δημιουργήθηκαν οι κανόνε παιχνιδιού και αυτό είναι πολύ σημαντικό ε, γιατί δεν ε, έχουν όλοι τα ωφέλη που θα έπρεπε στην ανάπτυξη δραστηριοτήτων σε αυτόν τον τομέα. Θα πρέπει επίση η αυξημένη χρήση πόρων να εξεταστεί και από τη σκοπιά τη εξάρτησή μα από την ενέργεια. Πρέπει να κοιτάξουμε προ Ανατολά για να καταλάβουμε πόσο σοβαρό είναι το θέμα αυτό. Και από την άποψη τη απόδοση των επενδύσεων και των, του κόστου που θα έχει αποφευθεί, ξέρουμε ότι τα υγειονομικά συστήματα ε, πιέζονται από, από του περιβαλλοντικού κινδύνου. Η βιοπικιλότητα και η απώλεια κεφαλαίων είναι στοιχεία που ε, επιφέρουν κοινωνικό κόστο. Η αναχέτηση και η προσαρμογή ω προ τι κλιματικέ αλλαγέ και το κόστος που θα αποφύγουμε εκεί είναι πολύ σημαντικά στοιχεία. Μια πρόσφατη μελέτη που δημοσιεύτηκε την περασμένη εβδομάδα από το Ερμένο Βασίλειο δείχνει ότι κάθε ε, λίρα που ξοδεύεται για περιβαλλοντικούς κανονισμούς και τη συμμόρφωση με αυτούς καθώς και το κόστος για τις επιχειρήσεις δίνει απόδοση περίπου τρει λίρες για κάθε μία λίρα. Επόμενη διαφάνεια. Ένα παράδειγμα του που η καινοτομία μπορεί να οδηγήσει σε πρωτοπόρες λύσεις και που είναι στην αιχμή της τεχνολογίας η Ευρώπη. Στα πράσινα τμήματα βλέπετε τις ε, επενδύσει για τη χρηματοδότηση της μετάβασης για το συνδυασμό ε, δημόσιων και ιδιωτικών κεφαλαίων. Από το 2007 η ΕΤΕ ανέλαβε ηγετικό ρόλο. Σε μία επταετία είδαμε η αγορά αυτή να αυξάνεται από το 1 δις ευρώ σε περισσότερα από 100 δις με την Ευρώπη να βρίσκεται πραγματικά σε πρωταγωνιστικό ρόλο. Ε, εν είδη συμπεράσματο, λοιπόν, πρέπει να πω ότι πιστεύουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 5 του προτινόμενου κανονισμού υπάρχουν πολύ σοβαροί λόγοι ω προ τι οικονομικέ επιδόσει, την απασχόληση και την ανταγωνιστικότητα, αλλά και ω προ την περιβαλλοντική πρόοδο να επικεντρωθούμε όντω σε ε, σοβαρέ λύσει στην πράσινη και κυκλική οικονομία στην Ευρώπη. Ευχαριστώ. Thank you very much. Ευχαριστούμε πολύ. Και περνάμε στον επόμενο μιλητή, που είναι ο Χωσέ Μαρία Μπάτ, που είναι επικεφαλής οικονομολόγος της Εθνικής Τράπεζας Πρόθεσης στην Ισπανία. Ευχαριστώ πολύ κύριε Αρτουή και κύριε Γκουαλτιέρη, αξιότιμοι ευρωβουλευτές, κυρίες και κύριοι. Πρώτα απ' όλα ευχαριστώ πολύ την Επιτροπή Προπολογισμών και την ε, Οικονομική Επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που οργάνωσαν την ακρόαση αυτή από κοινού. Και σας ευχαριστώ φυσικά που με προσκαλέσατε. Μετά από 8 χρόνια, μετά από την αρχή της κρίσης, τώρα αρχίζουν οι επενδύσεις. Σύμφωνα με το οι εκτιμήσεις σήμερα είναι 280 δισεκατομμύρια, 170 θα είναι στον οικοδομικό τομέα. Τι σημαίνουν αυτές οι εξελίξεις. Από τη μια μεριά υπάρχει μια σύμμετρη σχέση όσον αφορά τις δημόσιες επενδύσεις. Οι κυβερνήσεις φυσικά περνάνε από μία περίοδο δημοσιονομικής λιτότητας και από την άλλη μεριά το Σύμφωνο Σταθερότητας έχει επηρεάσει τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, έχουν γίνει πιο ευάλωτες. Το επενδυτικό αυτό πρόγραμμα λοιπόν από το 2014 που μας ανακοίνωσε ο κύριος Γιούγκερ και ονομάζεται Γιούγκερ επενδυτικό πρόγραμμα σίγουρα θα προωθήσει τις επενδύσεις στις μεταφορές και στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Οι εγγύσεις θα επιτρέψουν την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων σε συνεργασία με τις Εθνικές Τράπεζες Πρόθεσης να αναλάβουν κινδύνους με νέα σχέδια, νέα έργα και να λειτουργήσουν καταλυτικά προκειμένου να επιτευχθεί η μόχλευση επί 15. Φυσικά θα υπάρξουν θετικές επιπτώσεις μακροπρόθεσμα. Προς το παρόν έχουμε τον ε, πολλαπλασιαστή τύπου Keynes και βάσει αυτού γίνονται οι υπολογισμοί Η απασχόληση φυσικά είχε πληγεί πάρα πολύ και το βασικό κριτήριο, βασική προϋπόθεση είναι να μειωθεί η ανεργία η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα διατηρήσει στα ίδια επίπεδα τους δείκτες της. Αυτό που είναι πιο σημαντικό λοιπόν είναι οι επενδύσεις και μακροπρόθεσμα και βραχυπρόθεσμα. Πρέπει να ερμηνευτούν σαν μια ικανότητα παραγωγική και θα πρέπει να ενισχύσει και την δυνατότητα των επενδύσεων αυτών να χρηματοδοτήσουν το δημόσιο χρέος σε πολλές χώρες. Για να μπορέσει να βελτιωθεί λοιπόν η κατάσταση και να ερμηνευτούν όλες αυτές οι επενδύσεις σε παραγωγή, πρέπει να υπάρξουν οι σωστές πρακτικές ομοιογενώς σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αποτελεσματικότητα και να αποφευθούν κίνδυνοι που έχουν να κάνουν με το δημοσιονομικό κόστος των αποφάσεων. Το επενδυτικό σχέδιο Juncker το φροντίζει αυτό. Παρόλο που επικεντρώνεται στην δημιουργία του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων, έχει υπόψη και πολύ πιο μακροχρόνιες προοπτικές. Το θέμα της επιλογής των έργων σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο συμπληρώνονται με την τεχνική αρρωγή που προσφέρει ένας συμβουλευτικός επενδυτικός κόμβος και θα βοηθήσει έτσι να υπάρχει μεγαλύτερη ομοιογένεια σε ολόκληρη την Ευρώπη. Βελτιώνεται επίσης το επενδυτικό πλαίσιο στην Ευρώπη, άρονται τα εμπόδια. Και αυτό φυσικά είναι ευπρόσδεκτο. Η δημιουργία του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων μαζί με τους διάλους πυλώνες του προγράμματος αποτελούν ένα μεγάλο βήμα προς τα μπρος για τις μεταφορές, για την καινοτομία, όπως έγινε και στι Ηνωμένε Πολιτείες. Έτσι θα υπάρξει επιμονή μου βάσεως ένας αντίκτυπος και στην Ευρώπη. Η Ευρώπη αντιμετωπίζει μια παράδοξη κατάσταση σήμερα. Δεν έχει επενδύσεις, ούτε βραχυπρόθεσμα, ούτε μακροπρόθεσμα. Γι' αυτό δύο πράγματα πρέπει να ληφθούν υπόψη προκειμένου να αντιμετωπίσουμε την ε, έλλειψη των επενδύσεων και να λειτουργήσει ικανοποιητικά το έτσι. Οι επενδύσεις πρέπει να γίνουν σε προγράμματα της διευκόλυνσης συνδέοντας την Ευρώπη εν ώψη του 2020. Ο πολυπλησιαστής εκεί είναι πολύ μεγάλος. Οι επενδύσεις αυτές ε, μπορεί να πετύχουν ακόμα μεγαλύτερο πολλαπλασιαστή. Δεύτερον, Τόλο όλο και με περισσότερα έργα τα οποία θα γραμματοδοτηθούν θα βελτιώσουν και τη διαδικασία επιλογής και θα αρούν διάφορους φραγμούς και εμπόδια αριθμιστικούς και άλλους που εμποδίζουν αυτή τη στιγμή τις εξελίξεις. Ο συνδυασμό λοιπόν αυτών των παραγόντων θα έχει σαν αποτέλεσμα εκθετικά να αυξηθεί ο πολλαπλασιαστής και να πολλαπλασιάσει ακόμα περισσότερο τα ποσά. Θα διασφαλίσουμε επίση συνεχείς βελτιώσεις και όσον αφορά την ποιότητα και όσον αφορά την ποσότητα. Η ανάγκη για επενδύσεις στην Ευρώπη είναι πολύ μεγάλη. Αλλά εδώ πρέπει να λάβουμε υπόψη μας τρεις διαστάσεις. Η πρώτη είναι ότι δεν υπάρχουν αρκετές ταπάνες στις διάφορες χώρες. Δηλαδή θέλω να πω ότι οι ανάγκες για επενδύσεις δεν συνδυάζονται με νέες υποδομές, αλλά με τη διατήρηση παλιών υποδομών που ήδη υπάρχουν. Οπότε η συντήρηση δεν έχει τα αποτελέσματα που θέλουμε για βιωσιμότητα και για χρήση του ιδιωτικού κεφαλαίου. Δεύτερη διάσταση. Ενώ οι επενδύσεις βέβαια μπορούν να υπολογιστούν εύκολα, Η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται πίσω σε σχέση με τις Ηνωμένες Πολιτείες, για παράδειγμα. Τεχνολογίες, ε, ε, ψηφιακά, τέτοιου είδους επενδύσεις είναι αναγκαίο να γίνουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το μείγμα ανάμεσα στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τις νέες ανάγκες για επενδύσεις διαφέρει βέβαια από χώρα σε χώρα στη Γερμανία πολύ περισσότερο από ό,τι στην Ισπανία. Και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να υπάρχουν και διαρθρωτικές αλλαγές στις συνθήκες επενδύσεων. Μια στρατηγική ενός μοντέλου για όλους πρέπει να αποφευθεί. Είναι σαφές ότι οι επενδύσεις από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Σταυγικών Επενδύσεων θα γίνουν με τέτοιο τρόπο που θα διαφέρει η κατάσταση από χώρα σε χώρα. Αυτό είναι σίγουρο και είναι λογικό. Μπορεί όμως να ερμηνευθεί σαν αδυναμία. Χρειάζεται μια καλή ισορροπία ανάμεσα σε νέα έργα και σε έργα συντήρησης, και ανάμεσα στις υλικέ και στις άειλες επενδύσεις. Έρχομαι τώρα στα τελευταία μου σημεία. Πρώτα απ' όλα, ο πολλαπλασιαστής των επενδύσεων του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων θα είναι κάτι θετικό. Δεύτερον, πρέπει να αυξάνονται συνεχώς τα επενδυτικά προγράμματα, αλλά να βελτιώνεται και η ποιότητά τους το πρόγραμμα αυτό μπορεί να έχει θετικές επιπτώσεις στις επενδύσεις έτσι κι αλλιώς και να έχει μακροχρόνιες επιπτώσεις, κάτι που είναι πολύ πιο σημαντικό από οποιοδήποτε πολλαπλασιαστή. Και τέλος, παρόλο που δεν υπάρχουν αρκετές επενδύσεις στην Ευρώπη, οι ανάγκες διαφέρουν από χώρα σε χώρα. Ευχαριστώ πολύ. Ο πρόεδρος Γκουαλτιέρη, σας ευχαριστώ πολύ κύριε. Τελευταίος ομιλητής για το πρώτο αυτό τμήμα, ο κύριος Χόλαντ, καθηγητής στην Οικονομική Σχολή του Πανεπιστημίου της Κουίμπρα. Έχει το λόγο κύριε. Ευχαριστώ. Εγώ διαφωνώ. Και μάλιστα ουσιοδός κατά τη γνώμη μου, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων αποτελεί εσφαλμένη αφετηρία για οποιαδήποτε ανάκαμψη. Δεν είναι αναγκαίο, δεν είναι βιώσιμο, δεν είναι χρήσιμο και με την έννοια μάλιστα ότι παραπλανά, διότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει όργανα που δεν βασίζονται στο εθνικό χρέος, δεν χρειάζονται ούτε εγγυήσεις από θεσμικά όργανα, ούτε από πουθενά. Τα έχω βάλει και σε ένα εγγραφό που ελπίζω ότι τα έχετε διαβάσει εσείς οι ευρωβουλευτές. Έχει τέσσερα βασικά στοιχεία το εγγραφό αυτό. Πρώτο, η πρόταση για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στατικών Επενδύσεων προέρχεται από μια έξοχη ανάλυση που έκανε ο Πολωνός Υπουργός Οικονομικών Σούρεκ για την ανάγκη μια ανάκαμψης στην ευρωπαϊκή οικονομία βασισμένη στι επενδύσεις. Όμως βασίζεται σε μια ασφαλμένη αντίληψη ότι το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων το οποίο ήδη υπάρχει και το οποίο εγώ είχα συστήσει το 1993 στον Ζακ Ντελόρ και αυτός το ίδρυσε το 1994 σύμφωνα με τον ε, κύριο Σούρεκ λοιπόν δεν μπορεί να προωθήσει την ανάκαμψη στη βάση των επενδύσεων. Ενώ αυτό το EFI ακριβώς αυτό το σκόπο είχε και το καταστατικό του του επιτρέπει να εκδίδει ομόλογα που δεν μπορεί η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων να εκδώσει και ούτε χρειάζεται. Και ούτε χρειάζεται να βασίζεται σε δημόσιο χρέο. Δεύτερον, τα κριτήρια για την ε, ανάκαμψη βασισμένη σε επενδύσει δεν χρειάζεται να σχεδιαστούν εκ, του, εκ μηδενός. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του ΕΣΕΝ του 1994 είχε συμφωνήσει να χρηματοδοτήσει τα διευρωπαϊκά δίκτυα μεταξύ αυτών και το ευρύ φάσμα. Το πρόγραμμα του 1997 ειδική δράσης του Άμστερνταμ δηλαδή επέκτηνε τις αρμοδιότητες Ευρωπαϊκής Τράπεζα Επενδύσεων έτσι ώστε να μπορεί να επενδύσει σε υγεία, εκπαίδευση, αστική ανα, αναζωογόνηση, πράσινες τεχνολογίες, περιβάλλον κλπ. και υποστήριξη μικρών και μεσών επιχειρήσεων. Με την έκδοση ομολόγων που ήταν και ένας από τους αρχικούς στόχους στις συστάσεις που είχα κάνει στον Δελόρ τότε. Ότι να μπορεί να χρηματοδοτεί δηλαδή ένα Capital Venture Fund, το AFI. Τρίτο, καταρχήν, το προτινόμενο Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων είναι PPP, δηλαδή κοινοπραξία ιδιωτικού και δημόσιο τομέα. Όπως ήδη, έχει διαπιστώσει ο Ματέο Σούρεκ, δεν έχει δημόσια χρήματα. Μάλιστα αναμένεται μόχλευση παράγοντα 15 και όπως λέει ο ίδιος ο Γιούργη Κατάινεν είναι υπερβολικά υψηλό αυτό. Αυτός λέει ο Κατάινεν δηλαδή ότι θα πρέπει να μειωθεί στο 5 αλλά και αυτό είναι πάρα πολύ υψηλό. Η αναλογία αυτή δεν πληρεί τις συστάσεις του Jean-Claude Juncker την ομιλία του που απίφθινε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πέρσι τον Ιούλιο για μια ανάκαμψη βασισμένη σε επενδύσεις και που θα χρηματοδοτείται από ομόλογα της ΕΤΕ ύψους 300 δισεκατομμυρίων. Έτσι λοιπόν το EFSI είναι talk shop και όχι workshop, δηλαδή κουβέντες. Αυτό που χρειάζεται η Ευρώπη είναι μια ανάκαμψη τώρα. Ποιος θα αποφασίσει και πότε και πώς. Ήδη έχουμε έχουν περάσει 8 μήνες από την έγκριση και τον διορισμό του Ζαν Κλοντ γιουνκερ στην επικεφαλής Ευρωπαϊκής Επιτροπής από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που εμένα με καταχαροποίησε. Αλλά τι λέω εγώ τώρα, εγώ λέω, μάλλον δεν λέω ότι πρέπει να ξεχαστεί το Ευρωπαϊκό Σύμφωνο Στατικών Επενδύσεων, αλλά θα πρέπει να αναγνωρίσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ελπίζω να το κάνει αυτό στην έκθεση που θα υποβάλει, ότι στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων. Με αυτά τα δύο δηλαδή υπάρχουν επαρκή εργαλεία για μια ανάκαμψη βασισμένη σε επενδύσεις, χωρί δημοσιονομικέ μεταφορές, χωρί δημιουργία νέων θεσμών και ιδίω χωρί εγγύσει. Όταν ο Πολωνός Υπουργός Οικονομικών Ματέο Ζούρεκ είπε ότι χρειάζεται το νέο Ευρωπαϊκό Ταμείο απευθυνόμενο στον Μπρούγκελ πέρσι τον Σεπτέμβρη, είπε ότι το μέγεθος του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων είναι μεγαλύτερο γιατί έχει το AFI, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων, μόνο 4,5 δισεκατομμύρια. Όμως πρόκειται για λάθος ανάγνωση της ιστοσελίδας. Το ίδιο το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων λέει ότι το 2.1, το άρθρο 2.1 προβλέπει ότι τα χρήματά του διατίθεται στην προώθηση κοινοτικών στόχων. Εγώ είχα πει ήδη τότε στον Τελόρ να χρησιμοποιηθεί ως το δυνατόν ευρύτερα. Δεν υπάρχει καμιά αναφορά στους κανονισμούς του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων ότι περιορίζεται μοναχά σε χρηματοδοτική υποστήριξη μικρών και μισών επιχειρήσεων. Το άρθρο 2.2 λέει οι δραστηριότητες του Ταμείου μπορούν να περιλαμβάνουν και επιχειρήσεις δανεισμού, δηλαδή επιτρέπει την έκδοση ομολόγων, και αυτό έχει επιβεβαιωθεί και από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων το 2012, σε έγγραφό της προς την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, ότι μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ανάκαμψη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεύτερο, υπάρχει το μέγα θέμα από πού θα προέλθουν τα χρήματα. Λένε πολλοί από τη Γερμανία, μα δεν χρειάζεται να προέλθει από πουθενά από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μπορούν να ανακυκλωθούν παγκόσμια πλεονάσματα. Είναι τεράστια δικλίμακα αυτών των παγκόσμιων πλεονασμάτων. Ο επικεφαλής του ΠΙΜΚΟ που είναι ε, μεγάλο ε, σταξιωτικό ταμείο είπε ότι θέλει να επενδύσει το ταμείο σε υψηλές αποδόσεις Επίσης, το Κινέζικο Ταμείο CIC έχασε το 2012 χρηματοδοτώντας δημόσιες επενδύσεις στην Ευρώπη και είπε ότι θέλει ομόλογα τουλάχιστον δεκαετούς αποδόσεως. Εγώ γνωρίζει ο Φίλιπ Μάιστα, τον εκτιμώ πάρα πολύ και ήταν πολύ χρήσιμη η συνάντηση που είχαμε το Δεκέμβριο εδώ στις Βρυξέλλες όταν σήκωσα το χέρι μου και είπα Μάλλον είπα εγώ, σηκώστε το χέρι σας όπου, όσοι από εσά γνωρίζετε ότι η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, τα δάνεια που δίνει, δίνει δηλαδή, δεν συνυπολογίζονται στο εθνικό δημόσιο χρέος. Όλοι τον εγνώρισαν αυτό. Και ο Φιλίπ Μέιστα το επιβεβαίωσε. Βεβαίω και έχει δίκιο να ανησυχεί ότι η Ευρωπαϊκή Τραπέζα Επενδύσεων ανησυχεί για την βαθμολόγησή τη τριπλού Α, διότι εξαρτάται η χρηματοδότησή τη από τα συνταξιοδοτικά ταμεία. Γιατί τα συνταξιοδοτικά ταμεία πάλι θέλουν οπωσδήποτε το τριπλό α της τράπεζας. Αυτό που μπορεί να γίνει όμως είναι το EFSI να ενισχύσει την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων προσελκύοντας χρήματα από τα παγκόσμια πλεονάσματα που πρόκειται για εκατοντάδες δισεκατομμυρίων και αυτό μπορεί να γίνει χωρίς καμιά ιδιαίτερη αύξηση στο καλυφθέν κεφαλαίο του. Υπάρχει μια διάκριση που είναι σημαντικό να γίνει μεταξύ της λέξης μόχλευση και της λέξης πολλαπλασιαστή μόχλευση σημαίνει μια αναμενόμενη, ένα αναμενόμενο πολλαπλασιασμό, αλλά δεν είναι πολλαπλασιαστή. Μια επένδυση που πολλαπλασιάζεται δημιουργεί πόρους. Το εφέ πολλαπλασιασμού της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων είναι μεταξύ 2,5 και 3, 3 φορές. Βάζοντας λοιπόν 100 δισεκατομμύρια, ανακυκλώνοντας πλεονάσματα από παγκόσμια συνταξιδοτικά ταμεία, μπορείς να πετύχεις τότε επί 2,5 ή επί 3 τα 300 δισεκατομμύρια στα οποία στοχεύει ο Ζαν Κλοντ Γιούνκερ και τα υποσχέθηκε ήδη από τον Ιούλιο στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και δεν νομίζω ότι θα πρέπει να τρομάζουν οι κυβερνήσεις από την στάση των οίκων αξιολογήσεων. Διότι έχει παραβλεφθεί για παράδειγμα τον Γενάρη του 2012 όταν η Standard και Poor μείωσαν την αξιολόγηση 9 χωρών μελών και έδωσαν τρεις λόγους, πρόσφεραν τρεις λόγους γι' αυτό. Αφενός η μείωση της μόχλευσης λόγω της περικοπής των δημοσίων προπολογισμών. δεύτερο, ότι δεν υπήρχε κανένα σχέδιο ανάκαμψης βασισμένο σε επένδυση. Χωρίς επενδύσεις δεν υπάρχει καμιά βιωσιμότητα για, τις, ε, για τα κρατικά ομόλογα και κατά τη γνώμη μου επίσης, και όχι μόνο κατά τη δική μου γνώμη βεβαίω, αλλά ε, θεωρώ ότι προκύπτει η πραγματικότητα, δεν χρειάζονται και νέα κριτήρια επενδύσεων φτιάξαμε ένα πάνελ για να συζητήσουμε τα πράγματα αυτά, δηλαδή στην ουσία κουβεντιάζουμε και ξανακουβεντιάζουμε αντί να λαμβάνουμε δράση. Ενώ το σχέδιο του Άμστερνταμ είχε ζητήσει από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων να χρηματοδοτήσει υγεία, εκπαίδευση, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις και μόνη της η αστική αναζωογόνηση, ανακαίνιση δηλαδή, μπορεί να σημάνει επενδύσεις σε κτίρια, σε συστήματα μετρό, ηλεκτρικού, ε, παροχή νερού κλπ. Και οικοδομές. Όλα αυτά είναι απολύτως βιώσιμα ήδη τώρα, χωρίς να χρειάζεται να περιμένει κανείς. Και θα πρέπει να ξεκινήσουν μάλιστα τα έργα αυτά, κατά τη γνώμη μου, κατά την άποψή μου, και όπως είχα συστήσει τότε στον Ζακ Τελόρ για, τη, για τη λευκή βίβλο του για τον ανταγωνισμό τότε, το 1993, όχι με νέα χρηματοδοτικά εργαλεία, τα οποία δεν τα δέχεται στο, στο κάτω της γραφής το ευρωπαϊκό κοινό. Βγείτε έξω και ρωτήστε ένα ταξιτζή τι γνώμη έχετε για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων. Δεν θα σας δώσει καμία συγκεκριμένη απάντηση. Αυτό που χρειάζεστε είναι ένα New Deal για την Ευρώπη. Όπως το New Deal του Roosevelt του 1930. Ο, New Roosevelt, ο, New, ο, Roosevelt ε, τότε πήρε τις αποταμιεύσεις και τις μετέφερε σε επένδυση και περιβαλλοντικού χαρακτήρα. βάλε η Authority για παράδειγμα. Αυτή ήταν η επιτυχία του. Μείωσε την ανεργία από 25 περίπου 100% σε κάτω του 10% μέσα σε 7 χρόνια πριν να ξεσπάσει βέβαια ο δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος. Και το έκανε αυτό με ομοσπονδιακό δημοσιονομικό έλλειμμα του 3%. Αυτά προβλέπει δηλαδή το όριο του Μάστριχτ. Σας προτείνω λοιπόν, σας συνιστώ προσοχή μην συνεχίζετε να μιλάτε και να μιλάτε και να μιλάτε ξανά για κάποιο νέο ταμείο. Αν θέλετε να μιλάτε, μιλάτε. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Αλλά στηρίξτε το γεγονός ότι ήδη υπάρχουν αυτοί οι δύο θεσμοί. Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων. Ανακυκλώστε τα παγκόσμια πλεονάσματα και βάλτε τα να δουλέψουν για την Ευρώπη. Και αυτό το Ευρωπαϊκό New Deal μπορεί να αρχίσει στους 8 μήνες τώρα. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε κύριε Χόλαντ. Όπως είδατε είχαμε ένα βρήφασμα απόψεων. Χρήσιμο αυτό. Και μαθαίνουμε ότι κατά την άποψη κάποιων το πρόγραμμα Juncker μπορεί να μην είναι ακριβώς αυτό που νομίζαμε. Τώρα να ακούσουμε τους εισηγητές μας για τη συνεισφορά τους ε, στη συζήτηση. Ο κύριος Μπούλμαν για τρία λεπτά ή ο κύριος Φερνάντες. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Να χαιρετήσω όλους τους προσκεκλημένους σε αυτό το πάνελ και χαίρομαι και για τη διαφορά απόψεων που ακούσαμε να υπάρχει. Εγώ είμαι από αυτούς που θεωρούν ότι το πρόγραμμα Juncker, αυτό το ταμείο, θα επιτρέψει πέραν των επενδύσεων, όπως ακούστηκε, θα επιτρέψει να περιοριστεί η γραφειοκρατία, να εμβαθύνουμε στην εσωτερική αγορά και όπως επίσης υπόθηκε να, στηρίξει, να στηρίξουμε τις επιχειρήσεις, ιδίως τις μικρομεσαίες. Πρόκειται για ένα εργαλείο επιπλέον που δεν ε, αμφισβητεί την αξία των υπόλοιπων εργαλείων και οργάνων που διαθέτουμε. Είναι συμπληρωματικό. Δεν θα υποκαταστήσει αυτά που ήδη υπάρχουν. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα πρέπει, μάλλον αυτό δεν σημαίνει ότι θα χάσουμε λοιπόν με το πρόγραμμα, αλλά θα κερδίσουμε. Ας ε, μην ξεχνάμε τον Καμίλου Μπράνκου Δεκαστέλου, έναν μεγάλο πορτοκαλοποιητή μετά τον Καμόη, ο οποίος έλεγε πάντοτε την εποχή των ανακαλύψεων οι Πορτογάλοι δεν ήξεραν τι θα πετύχουν, έφευγαν τα καράβια για να ανακαλύψουν ένα νέο κόσμο, αλλά δεν το γνώριζαν εκ των προτέρων. Αυτό λοιπόν είναι ο δικός μας ρόλος. Έχουμε ακόμη κόσμους ολόκληρους μπροστά μας να, καλύψουμε. Υπάρχουν ιδιωτικά ε, προγράμματα και έργα που μπορούν να εκτελεστούν, να διευκολυνθούν και να δημιουργήσουν θέσεις απασχόλησης αλλά και ανάπτυξη. Θα αναφέρω τώρα μια ερώτηση, μια ανησυχία δική μου ή των επενδύσεων θα κάνει ένα είδος προεπιλογής το λεγόμενο κομιτέ ντανδεστισμό. Μετά όμως θα αποφασίζει η ΕΤΕ. Η επιλογή και η ευελιξία της επιλογής είναι κάτι που θα κορίστηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτή τη διαδικασία προβλέψαμε. Θα πρέπει να την αποσαφηνίσουμε όμως πώς ακριβώς θα λειτουργεί. Και επίσης η ανάγκη συνοχής. Εδώ έχουμε ένα πρόγραμμα που θα πρέπει να καλύψει ελλείψεις της αγοράς. Αυτό θα πρέπει να γίνει σαφές. Υπ' αυτήν την έννοια η πλατφόρμα επενδύσεων που έχει σχεδιαστεί που την αναφέρατε και εσείς, θα διαρθρώσει τα διάφορα έργα μια πλατφόρμα που πιστεύω ότι θα πρέπει να είναι δωρεάν στη χρήση της για να επιτρέψει ακριβώς να υπάρχουν οι απαραίτητες ζυμώσεις για την εδαφική συνοχή με τα κενά στην αγορά που θα πρέπει να έρθει να καλύψει ακριβώς το πρόγραμμα. αυτή η βοήθεια διάρθρωση των προγραμμάτων με την πλατφόρμα επενδύσεων που θα συναρθρώσουμε στο όλο εγχείρημα, νομίζω ότι είναι μια πολύ σημαντική διάσταση του προγράμματο αυτού. Ευχαριστώ. Econ Ούντο Μπούλμαν, εισηγητής της Επιτροπής Οικονομικών, ΕΚΟΝ. Ευχαριστώ και εσά, κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ και εσά, κύριε Εμπειρογνώμονε. Βρίσκω ότι αυτή η συζήτηση που διεξάγουμε σήμερα έχει χαρακτήρα πραγματικά δυναμικό είναι μάλιστα πολύ ενδιαφέρουσε και οι παρεμβάσει και ελπίζω να γίνουν ενδιαφέρουσε ερωτήσει. Ήταν πραγματικά φρέσκια ανάσα η παρέμβαση του Στουαρτ Χόλαντ. Ερώτηση. Το Κοινοβούλιο. Δεν είναι εκείνο ο οποίο λέει τελικά τι θα γίνει. Και εγώ εκφράζω τη λύπη μου γι' αυτό και την έχω εκφράσει και άλλε φορέ. Ούτε μπορούμε να πούμε στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων τι θα κάνει. Και αυτό με ναι. λυπεί και εκφράζω τη λύπη μου αυτή. Ακόμα περισσότερο δεν λυπούμε που ούτε καν στις χώρες μέλη δεν μπορούμε να πούμε τι να κάνουν. Έχουμε λοιπόν μπροστά μα αυτό το προϊόν και πρέπει να το διαμορφώσουμε. Λέτε εσεί ότι δεν επιθυμείτε να καταργηθεί. Άρα πρέπει να εξετάσουμε τι θα πρέπει να ή τι θέλουμε να αλλάξει στο προϊόν αυτό εντό εισαγωγικών. Ρωτώ λοιπόν για να μου δώσετε κάποιε πιο συγκεκριμένε. ιδέε με εμπνέει η παρέμβαση του κύριου Μάιστατ. Συμφωνώ μαζί του σε ορισμένα σημεία και έχω και ερωτήσεις. Εκτός από τη γενική παρατήρηση βρίσκω σωστό αυτό που λέτε ότι χρειάζεται κοινοβουλευτικός έλεγχος που θα στρέφεται ιδίως στην Διευθυντική Επιτροπή σε ό,τι αφορά τη χρηματοδότηση, την συγχρηματοδότηση των χωρών μελών. Αυτή να λειτουργήσει με λογικό τρόπο και σε αυτό συμφωνώ. Ερώτηση. Πώς μπορεί να φροντίσει κανείς ώστε με τα νέα μέσα να μπορούν, εννοείται χρηματοδοτικά μέσα, να μπορούν να αναλυφθούν πιο, μάλλον επενδύσεις μεγαλύτερου κινδύνου. Πώς μπορεί δέκα να συμβάλλει κανείς, ώστε οι επενδύσεις να κατευθυνθούν, για παράδειγμα, περισσότερο σε τομείς που θεωρεί πιο σημαντικούς ο κ. Μπράινγκς, και στο οποίο συμφωνούμε ορισμένοι από εμά. Η τάση για επενδύσεις δηλαδή του νέου ταμείου να οδηγήσει την επένδυση, μάλλον τη χρηματοδότηση σε επενδύσεις που δεν τις πολύ θέλουν ακόμα. Για μας αυτό αποτελεί ένα είδος μαύρου κουτιού και πρέπει να ανοίξει. Δεύτερη ερώτηση το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων να συνεχίσει απλά αυτά που κάνει υπέρ των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων που ούτως ή άλλως κάνει μέχρι τώρα. Αυτό δεν μπορεί να αρκεί. Πώς λοιπόν θα μπορέσουμε να διαμορφώσουμε μια στρατηγική που να βοηθήσει περισσότερο τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Βέβαια τελικά οι τράπεζες και πάλι θα αποφασίσουν πού θα δώσουν τις πιστώσεις και πώς θα κρίνουν τους κινδύνους. Δεν έχουμε καμιά επιρροή εμείς στο πώς μπορούμε να βοηθήσουμε περισσότερο τις μικρομεσαίε επιχειρήσει με τον τρόπο αυτό. Κυρία Αμπάντ, πού βλέπετε τη δυνατότητα να μπει μια εθνική τράπεζα επενδύσεων που έχει κάποιο ρόλο. Πού μπορεί να ενταχθεί μέσα σε μια νέα στρατηγική του EFSI αυτή, αυτού του είδους η τράπεζα, ε, της οποίας συνηγορήσατε και εσείς. Μάλιστα, ευχαριστώ. Κύριος Μάιστατ. Παρακαλώ, δύο λεπτά. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα απαντήσω και στον κύριο Φερνάντες και στον κύριο Μπούλμαν στην πρώτη του ερώτηση. Έχει να κάνει με τον ρόλο της Επιτροπής Επενδύσεων. Δεν είναι η Επιτροπή Επενδύσεων εκείνη η οποία θα προεπιλέγει τα έργα. Εξάλλου τα κείμενα εξελίχθηκαν. Στην πρώτη εκδοχή του κανονισμού όντως ήταν ε, ένα καθήκον που είχε ανατεθεί σε αυτή την Επιτροπή. Σφάλμα όμως, γιατί δεν γίνεται. Πώς θέλετε έξι εμπειρογνώμονε που δεν είναι και full time, ακόμα και αν είναι αρμόδιοι, να μπορούν να επιλέξουν από τα εκατοντάδε ε, προγράμματα, έργα που έχουν υποβληθεί από τις χώρες μέλη. Πρόκειται για ένα τεχνικό έργο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων που μπορεί να το κάνει, που είναι εξοπλισμένη γι' αυτό και που μπορεί να προσλάβει και επιπλέον προσωπικό. Η Επιτροπή λοιπόν Επενδύσεων στην τελευταία εκδοχή τουλάχιστον θα κοιτάει τα έργα τα οποία έχουν προεπιλεχθεί από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων θα καλύπτουν τις προϋποθέσεις που προβλέπονται από τον κανονισμό, το άρθρο 5. Και από τους, τις κατευθυντήριες γραμμές ε, της ε, Επιτροπής Κατεύθυνσης. Πρέπει λοιπόν να διασφαλίσουμε, κύριε Μπουλμαν, ότι η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων θα μπορέσει έτσι να χρηματοδοτήσει τα έργα υψηλότερου κινδύνου, που αλλιώς δεν θα χρηματοδοτούντουσαν. Αυτό είναι ο ρόλος της Επιτροπής Επενδύσεων, να διασφαλίσει ότι συνάδουν με τον κανονισμό βάσει της ανάληψης κινδύνου έτσι όπως προβλέπετε. Αυτό θα ελέγχει η Επιτροπή Επενδύσεων. Αν διαπιστωθεί ότι το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικής Επενδύσεων έτσι κι αλλιώς χρησιμοποιείται για έργα τα οποία έτσι κι θα μπορούσαν να είχαν επενδυθεί, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, είναι περιττό. Τα ατομικά έργα η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων λοιπόν μπορεί καλύτερα να τα εκτιμήσει και να δούμε κατά πόσο τηρούνται οι προσανατολισμοί της Ευρωπαϊκής Επιτροπής υπό τον έλεγχο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα κάνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και αυτή η Πιλωτική Επιτροπή. Για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις τώρα. Ο πρόεδρος μου λέει ότι φτάνει. Δύο λόγια γι' αυτό. Μέχρι τώρα δεν είδα τίποτα πραγματικά καινούργιο για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Όταν διαβάζετε το κείμενο, και τουλάχιστον έτσι το αντιλαμβανόμαστε και το αντιλαμβάνετε και το ΕΦΕΗ, είναι για να κάνει κάτι παραπάνω από ό,τι γίνεται μέχρι τώρα. Δηλαδή να στηρίξει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις είτε μέσω εγγυήσεων στις τράπεζες οι οποίες δανείζουν τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις ή μέσω κεφάλαιων, κεφαλαίων κινδύνου που επενδύονται. Ακριβώς για να μπορούν να κάνουν κάτι παραπάνω, όχι όμως κάτι διαφορετικό. Ευχαριστώ. Ο κύριος Μπρίνιξ έχει τώρα τον λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα προσπαθήσω να είμαι σύντομος. Τα κριτήρια αυτά, πώς μπορεί κανείς να τα πάρει σοβαρά, ρωτήσατε. Θέλω να απαντήσω τρία πράγματα. Πρώτον, παίρνοντας σοβαρά τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις υποχρεώσεις που αναλαμβάνει. Προς το παρόν υπάρχουν χιλιάδες στόχοι και πακέτα πολιτικής στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν λοιπόν θέλετε πραγματικά να πετύχετε τους στόχους, αυτό πρέπει να γίνει. Δεύτερον, αν βασιστούμε σε αποδείξεις που έχουμε μέχρι τώρα, ότι όντως λειτουργούν αυτά και ότι όντως φέρνουν αποτελέσματα στην κοινωνία, όχι μόνο για το περιβάλλον, για το κλίμα, αλλά και για την οικονομία. Επίσης, λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 5 του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων, τρία από τα πέντε κριτήρια συνδέονται πολύ στενά με τους στόχους που προωθούμε. Στόχους έρευνας, ανάπτυξης που έχουν να κάνουν με τον Horizon 2020 για τα 20 δισεκατομμύρια ευρώ. Πολλά χρήματα που μπορούν να στηρίξουν το πακέτο. Και τρίτον, λέγοντας ότι όσον αφορά την, τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος, να ξέρω ότι έχουμε συζητήσει με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για το πώς μπορούμε να βελτιώσουμε τη στήριξη της τράπεζας για τέτοιου είδους επενδύσεις. Αυτά έχω να απαντήσω εγώ. Πρόεδρος, ευχαριστούμε. Κύριο Σάμπατα. Τρεις παρατηρήσεις από πλευράς μου. Πρώτα απ' όλα συμφωνώ απολύτως με τον κύριο Φερνάντες. Είπε ότι το ΕΦΣΥ δεν υποκαθιστά τα υπάρχοντα οχήματα και αυτό συμβαίνει γιατί ακριβώς δεν μπορεί. Το βασικό ταμείο μπορεί να δημιουργεί ένα πρόβλημα. Δεν μιλάμε όμω στην πραγματικότητα για ταμείο. Μιλάμε για μια εγγύηση που παρέχει η Ευρωπαϊκή Τράπεζα προ την ε, ε, ΕΤΕ. Δηλαδή είναι μια εγγύηση με τα υπάρχοντα οχήματα. Έτσι θα αναλάβουν περισσότερου κινδύνου η ΕΤΕ και οι Εθνικέ Τράπεζε. Αυτό είναι σημαντικό, διότι δεν υπάρχει κάτι νέο που δημιουργείται. Δεύτερον, ο κύριος Μπούλμαν ρώτησε τι μπορούμε να κάνουμε για να το, να το διασφαλίσουμε αυτό. Νομίζω ότι θα κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε. Δηλαδή να δημιουργήσουμε τα κατάλληλα κίνητρα εκ των προτέρων για το προσωπικό του ΕΦΣΥ και μετά να προβλέψουμε τα απαραίτητα συστήματα ε, εκ των υστέρων αξιολόγησης. Μόλις έχουμε αυτά τα δύο συστατικά, δηλαδή το να μάθει κανείς την πράξη, θα δείξει την αξία του οχήματο στην ε, πορεία του χρόνου. Αυτό μπορούμε να κάνουμε. Και τρίτο σημείο, ρωτήσατε τι μπορούν να κάνουν οι Εθνικές Τράπεζες Επενδύσεων. Εδώ μιλάμε για μια εγγύηση θα μπορεί να δώσει εγγυήσει προ τι εθνικέ τράπεζε στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Στατικών Επενδύσεων μέσω της ΕΤΕ. Στην ουσία είμαστε και εμεί τράπεζε με υπαγωγή στου ίδιου κανόνε που ισχύουν για τι τράπεζε. Θα δούμε τι ένταση, τι ισχύ μπορεί να ε, προκύψει και τι εγγύησει θα δεθούν μεμονωμένα στι επιμέρου χώρε και πολιτικός μέσω, των, ε, μέσω τη πλατφόρμα επενδύσεων. Ένα παράδειγμα θα μπορούσε να είναι το ε, πρόγραμμα των συγκεκριμένων επενδύσεων μέσω τη πανευρωπαϊκή πλατφόρμα. Stuart Holland. Ευχαριστώ για τα πρώτα αυτά σχόλιά σας. Κοιτάξτε, να το πω απλά. Ο Φιλίπ Μάιστατ είπε για την αξιολόγηση των έργων. Έξι εμπειρογνώμονες που δεν θα είναι καν full time και δεν θα μιλούν, θα μιλούν, θα μιλούν, θα μιλούν, μόνο αυτά κάνουν. Δεν είναι ταμείο, διότι δεν έχει χρήματα. Έχει μάλλον προφυλακτικό χαρακτήρα. Και στην ουσία αυτό που κάνει είναι να εμποδίζει το να μπορέσει να χρησιμοποιήσει, να βασιστεί μάλλον η ανάκαμψη στα εφιστάμενα εργαλεία. Ευχαριστούμε. Και τώρα στις ερωτήσεις και τις παρεμβάσεις των μελών. Πρώτος, η κυρία Γκάρτια Θαμπάλ, η της Επιτροπής Προπολογισμών. μισή λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα προσπαθήσω σε 1,5 λεπτό να συγκεντρώσω όλες τις ερωτήσεις και όλες τις αμφιβολίες που έχουν προκύψει κατά τη διάρκεια των εργασιών μας όσον αφορά το ταμείο αυτό. Εννοείται ότι ό,τι έχουμε το έχουμε μπροστά μας και μπορούμε να είμαστε επικριτικοί όχι, αλλά εν πάση περιπτώσει ο στόχος είναι να προσπαθήσουμε να βελτιώσουμε το σχέδιο, την πρόταση που μας κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δουλεύουμε λοιπόν πάνω στην εξή γραμμή. Θέλουμε να δούμε πώς μπορούμε να μειώσουμε τις μειώσεις του Europe Facility και του Horizon 2020. Μία από τις ιδέες λοιπόν που έχουμε για τη μείωση των επιπτώσεων αυτών είναι να βρούμε εναλλακτική χρηματοδότηση, να προσπαθήσουμε να χρηματοδοτήσουμε με περιθώριο από τον προϋπολογισμό, δημιουργώντας ε, το Ταμείο Εγγύσεων κλπ. Αλλά μια άλλη δυνατότητα και θα ήθελα να ξέρω από τον κύριο Μάιστατ ποια είναι η θέση του επ' αυτού. Πιστεύετε ότι μπορούμε να μειώσουμε το Ταμείο Εγγύσεων δηλαδή από τα 8 δις που μπλοκάρουμε στον προπολογισμό χωρίς να αγγίξουμε καθόλου τα 16 δις της εγγύησης. Πιστεύετε ότι αν μειώσουμε το ταμείο αυτό και βάζουμε σε, διακινδυνεύουμε τη συμμετοχή του ταμείου και τη λειτουργία του ταμείου αυτού. Και δεύτερον, Πιστεύετε πως είναι δυνατόν η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων να συμμετέχει με μεγαλύτερο κεφάλαιο, όχι μόνο με τα 5 δις δηλαδή, αλλά χρησιμοποιώντας ε, από θέματα πλεονάσματα μόνο που έχει από προηγούμενες χρονιές, ώστε να έχουμε στη διάθεσή μας περισσότερα χρήματα για το μέλλον. Πάρα πολλές παραπάνω ερωτήσεις θα μπορούσα να υποβάλω, αλλά θα περιοριστώ σε αυτές προς το παρόν. Ευχαριστούμε. Ο κύριος από την Επιτροπή Προπολογισμών. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να τονίσω και πάλι ότι από την άποψή μας δηλαδή των Ευρωπαίων συντηρητικών και μεθαρρυθμιστών έχω ακόμα πολλά ανοιχτά ερωτήματα για αυτό το Ταμείο Στατικών Επενδύσεων. Κρίσιμο είναι το εξή ερώτημα. Πού βρίσκεται όλη αυτή την αισιοδοξία ότι δηλαδή μπορείτε να λύσετε παλαιά προβλήματα με ένα νέο τρόπο. Δεν μπορώ δηλαδή να ειδώ πώς μπορεί να συγκεντρωθεί ένα τόσο μεγάλο ποσό για επενδύσεις χωρίς να ξέρουμε πού θα κατευθυνθούν, σε ποιες επενδύσεις βλέπω ένα καλάθι που θα μαζέψει χρήματα, δεν βλέπω κανένα καλάθι που να περιλαμβάνει, να έχει μέσα σχέδια επενδύσεων. Αυτά τα έχουμε ξαναδεί και ξέρουμε που οδήγησαν στην ιστορία. Πάνε τα κράτη να κατευθύνουν τις επενδύσεις. Ποιος αναλαμβάνει όμως την εγγύηση ότι θα είναι εξασφαλισμένη μακροπρόθεσμα η χρηματοδότησή τους. Τέτοια εγγύηση μπορεί να δώσει μονάχα η επιχείρηση, όχι το κράτος. Είναι απολύτως εσφαλμένη η κατεύθυνση και δεν αντιλαμβάνομαι την αναγκαιότητα. Αντιμετωπίζουμε μια πλημμυρίδα χρήματος, μηδενικά επιτόκια, δεν λείπουν λεφτά. Αυτά που λείπουν είναι σχέδια επενδύσεων και φοβούμε πάρα πολύ ότι πάμε να χρηματοδοτήσουμε επενδύσεις πάρα πολύ ψηλού κινδύνου. Ευχαριστώ. Ο κύριος Ότμαν Κάρας, Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε, κύριε και κύριοι. Επανέρχομαι σε αυτά που είπε ο Ούντο Μπούλμαν. Δεν πρόκειται εδώ για ευχολόγια, ούτε μόνο για αναλύσεις. Θα θέλαμε από... Χτυπάει το τηλέφωνο του κύριο Κάρας, δεν ακούμε τίποτα. Θα θέλαμε ο καθένας από τους εμπειρογνώμονε να κάνει μια συγκεκριμένη παρατήρηση για το σχέδιο της Κομισιόν. Δυστυχώ έχει τρομερέ παρεμβάσεις στο τηλέφωνό του. Ο Πρόεδρος, παρακαλώ επαναλάβετε γιατί δεν μπορούν να παρακολουθήσουν οι διερμηνεί. Θα ήθελα λοιπόν, λέει ο κ. Κάρα, κάθε ένα από του παρισταμένου εμπειρογνώμονε να μα εξηγήσει ακριβώς που θεωρεί ότι πρέπει να γίνει κάποια τροποποίηση στην πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Δηλαδή, τι θεωρεί ότι πρέπει να τροποποιηθεί έτσι ώστε να επιτευχθεί καλύτερο στόχος. Δεύτερο, ο κ. Μάιστατ είπε ότι με τα 16 δις δεν φαίνεται να είναι σίγουρο ότι μπορούν να προσελκύσουν περισσότερα χρήματα. Ερώτηση. Από πού πρέπει να προέλθουν τότε τα χρήματα έτσι ώστε η προστιθέμενη αξία αυτών των 16 δις να καταστεί καθαρή, σαφής και γι' αυτόν. Τρίτο. Είναι ορθό ότι το Ταμείο για το οποίο συζητούμε θα επιτύχει τους στόχους του μόνον εφόσον εγγράψουμε στον κανονισμό ότι δεν επιτρέπεται να, χρησιμο... να ε, χρηματοδοτήσει ούτε, ούτε ένα έργο το οποίο θα μπορούσε να χρηματοδοτηθεί από άλλα υφιστάμενα ταμεία. Πρόεδρος Γκουαλτιέρη, σας ευχαριστώ. Ο κύριος Ντεπρέ. Ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ και όλους τους ομιλητές για αυτή τη συζήτηση. Να τονίσω ότι όπως και ο κύριος Μάιστατ βρίσκω απαραίτητο αναγκαίο το πρόγραμμα αυτό και κυρίω στο πλαίσιο των μέτρων που ελήφθησαν από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Πρέπει να γίνει μια ομαλή μετάβαση. Ακούω συχνά να λέγεται ότι το πρόγραμμα αυτό θα βοηθήσει τι μικρομεσαίε επιχειρήσει. Όμω, αν δούμε του κανόνε, δεν βλέπω τίποτα συγκεκριμένο για τι μικρομεσαίε. Μιλούμε για επιχειρήσει μέχρι 3.000 εργαζομένου, μισθωτού. Ε, αυτό θα μπορούσε να είναι μια θεατρική τη ε, Google, τη Microsoft, οποιασδήποτε εταιρεία, αλλά δεν βλέπω τίποτα συγκεκριμένο για τι μικρομεσαίε. Θέλω λοιπόν να καταλάβω, ε, εάν το βλέπετε εσεί. Έπειτα, νομίζω ότι η ΕΤΕ θα τη βγάλει καθαρή από όλη αυτή την υπόθεση. Αν διαβάσετε του κανόνε, λέει ότι κάθε χρόνο θα λαμβάνει τουλάχιστον 20 εκατομμύρια ευρώ για την Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα Συμβουλών προ τι Επενδύσει. Αυτό λέει το άρθρο 2. Και δεύτερον, όπω θυμήσατε κύριε Μάιστατ, είναι η μόνη που θα υποφεληθεί από την εγγύηση. Επιπλέον, σε καθένα σε κάθε μια από τις περιπτώσεις των επενδύσεων θα, κατά, θα παρέμβει κατά ένα πέμπτο. Ε, εγγύηση κατά ένα πέμπτο και χρηματοδότηση του ενός πέμπτου από προγράμματα που θα πάρουμε κονδύλια όπως το Horizon 2020 ή το Connecting Europe Facility. Η ερώτησή μου λοιπόν είναι η εξή. Όλα αυτά για την ΕΤΕ, για έργα για τα οποία λέτε ότι η προστατικότητα δεν είναι εγγυημένη, δηλαδή θα πρέπει να ε, αναζητηθούν οι κατάλληλοι μηχανισμοί και καθώς θα υπόκειται ε, στις ανάγκες των χωρών, αλλά αυτό δεν το λέει. Ε, πουθενά στου κανόνε. Και επειδή μπορεί να συγκεντρωθούν οι επενδύσει σε συγκεκριμένε χώρε τελικά. Είναι πολλά τα στοιχεία, έτσι. Ε, άρα η ερώτησή μου είναι η εξή. Είναι απαραίτητο στην ε, σημερινή κατάσταση των πραγμάτων και ε, εφόσον θα πρέπει κάποιο να τροφοδοτήσουμε αυτό το ταμείο με τι εγγύσει, πρέπει από τώρα να πούμε πώ θα βρούμε αυτά τα οκτώ δι. Δεν μπορούμε απλώ να τα δώσουμε με μια πολιτική χειρονομία και να λέμε ότι κάθε χρόνο ανάλογα με ένα συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα που θα καθορίσουμε ε, με δόσει, ότι θα τα προβλέψουμε αυτά από το δημοσιονομικό πλαίσιο. ανάλογος με το που πρέπει να τα πάρουμε κάθε φορά για να ε, καλυφθεί το θέμα, το, η διάσταση των εγγύσεων. Νομίζω ότι για μα είναι σημαντικό να έχουμε μια εναλλακτική σε αυτό που θα ονομάσω άρθρα 18 και 19 τη πρόταση. Ευχαριστούμε. Η κυρία Ριάντα. Ευχαριστώ. Δεν προβλέπεται η γλώσσα της ομιλήτριας. Μιλεί, μιλεί κέλτικα η κυρία Ριάντ, τα οποία δεν γνωρίζουμε και θα περιμένουμε να δούμε αν θα μεταφραστούν από την συνεργάτηδά της. Sorry. Ε. Ο πρόεδρος Γκουαλτιέρη. Σύμφωνα με την εφαρμογή της αποφάσεως του προεδρίου δεν υπάρχει μετάφραση από την κελτική γλώσσα. Η κυρία Λυπούμε πολύ. Δεν μπορεί να γίνει. Δεν μπορεί ούτε να γίνει διαδοχική μετάφραση από την συνεργάτη δάσα σύμφωνα με τους κανόνες του Κοινοβουλίου. Ή θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε άλλη γλώσσα ή δεν, ή δεν θα σας επιτρέψω να αγορεύσετε συνεχίζει στα κερδικά. Ah, okay, so we move to the next speaker. Περνάμε στον επόμενο μιλητή, λέει ο Πρόεδρος, ο κύριος Τρεμόζα. Α, δεν είναι εδώ ο κύριος Τρεμόσα. Ο κύριος Δεμάτζη. Thank you, Chair. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πρώτα ευχαριστώ τους εμπειρογνώμονες για τις ε, παρεμβάσεις τους, ιδίως του κυρίου Χόλαντ, και η ομάδα της Ενωτικής Αριστεράς προτίθεται να μεταφέρει τις απόψεις του αυτές σε συγκεκριμένες τροπολογίες. Είναι πεπισμένη η πολιτική μου ομάδα ότι παρόλη την τεράστια ρευστότητα, παρά τους μηδενικούς ε, ρυθμού των επιτοκίων, δεν υπάρχει λόγος. Παρ' παρόλα αυτά βλέπουμε ότι έχουν καταρρεύσει οι ιδιωτικές επενδύσεις. It's the austerity stupid, θα έλεγα παραφράζοντας το It's the economy stupid του Πρόεδρου Κλίντον. Μάλιστα το ίδιο το ελεγκτικό συνέδριο της Ομοσπονδιακής Γερμανίας η, Ευρωπα... απάντηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που έδωσε μάλιστα και, στις... και στην... Ε, ερωτήσεις και απαντήσεις δίνει την προσπάθεια... κάνει την προσπάθεια αυτή διότι ακριβώς το χρέος είναι τόσο υψηλό και ο κύριος Τιούρα Τόλεντ είπε ότι θα ήταν δυνατό η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων να κάνει επενδύσεις χωρίς να βασίζεται καν στα κριτήρια του Μάστριχτ. Γι' αυτό ρωτώ πώς αιτιολογείται ότι για παράδειγμα εξαιρούνται οι ε, συγχρηματοδοτήσει των χωρών μελών, όχι όμως από, από τη ρήτρα δηλαδή του ορίου του Μάστριχτ. Thank you. Ευχαριστούμε. Εκ μέρους των Πρασίνων από την Επιτροπή Προπολογισμών, ποιος θα πάρει το λόγο. Ένας. Ο κύριος Τάραν. Ναι. Ευχαριστώ κύριε Γκουαλτιόρη. Δεν χρειάζεται να ρωτήσω τίποτα. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Ευτυχή. Ο κύριος Τζάνι έχει τώρα το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ τους ομιλητές διότι τελικώς μετά από εβδομάδες υποκριτικής τάσης και αδικαιολόγητου ενθουσιασμού για το πρόγραμμα αυτό αρχίζουμε να καταλαβαίνουμε πως το πρόγραμμα Juncker βασίζεται σε ε, υποθέσεις που δύσκολα θα ε, υλοποιηθούν και θα, γίνουν, θα λάβουν σάρκα και ωστά. Τρεις γρήγορες ερωτήσεις προς τους ομιλητές. Πρώτον, νομίζω, έχω την εντύπωση ότι στην ουσία έχετε μια μεγαλύτερη, σε μεγαλύτερη έκταση μετάφραση των ε, ομολόγων έργων της ΕΤΕ που δεν έχει δώσει ως τώρα καθόλου ε, ικανοποιητικά αποτελέσματα. Το πρώτο πρόγραμμα που χρηματοδοτήθηκε, το Κάστορ στην Ισπανία, ήταν ε, καταστροφή, διασπάθηση δημόσιων κονδυλίων. Ήθελα λοιπόν να καταλάβω, να μου πείτε τι γνώμη έχετε εσείς οι ομιλητές για, για αυτό το δικό μου το σχόλιο. Δεύτερη ερώτηση, η χρήση τις ε, κοινοπραξία ιδιωτικού δημόσιου τομέα. Είδαμε πολύ συχνά ότι το εργαλείο αυτό, η χρηματοδότηση έργων, δεν αποδίδει και μάλιστα ο κίνδυνος, αυτό που συνήθως συμβαίνει, είναι ότι γίνονται δημόσιες οι απώλειες από αυτό του είδους τα έργα και αν υπάρξουν ωφέλη κέρδη, αυτά ε, περνάνε στα χέρια των ιδιωτών. Ε, άρα, πώς θα μπορέσουμε να βρούμε εργαλεία εναλλακτικά για να μην χρησιμοποιήσουμε αυτή τη σύμπραξη ιδιωτικού δημόσιου τομέα που δεν έχει αποδειχθεί χρήσιμη. Ε, και ένα τρίτο σημείο, στο οποίο με συγχωρείτε, λέει ο Πρόεδρος, ε, πρέπει να κλείσετε. Ε, η ιδιωτικοποίηση δημόσιων υπηρεσιών, βασικών δημόσιων υπηρεσιών μέσα αυτό το ταμείο, Πώ μπορούμε να το παρεμποδίσουμε αυτό και πώ θα αντιμετωπίζετε εσεί αυτό το κίνδυνο. Ευχαριστούμε για του πράσινου ο κ. Έκχαουτ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Να συνεχίσουμε με τον παράγοντα πολλαπλασιαστή, αν και όπως είπαμε είναι καλύτερα να το λέμε μόχλευση. Επί 15 λέμε. Ανάμεσα σε αυτά που λέει ο κύριος Μάιστατ και ο κύριος Μπάξετ υπάρχει μια διαφορά. Γιατί αν αυτό το ταμείο πρέπει να μας βγάλει από το βάλτο εκεί που βρισκόμαστε, δεν πρόκειται για μια γνωστή κατάσταση, πρόκειται για κάτι καινούριο, πρόκειται για μια μετατροπή της οικονομίας. Αλλά αν δείτε την ε, σημερινή εμπειρία που έχουμε με τη μόχλευση όσον αφορά για παράδειγμα το Ταμείο για την Ενεργειακή Απόδοση, εκεί βλέπουμε μία μόχλευση 7. Οπότε το 15 δεν μπορεί να επιτευχθεί όταν προχωράμε σε πραγματικές ε, αλλαγές και τροποποίησεις. Πώς θα το πετύχουμε αν συνεχίσουμε να κάνουμε τα πράγματα όπως ξέραμε και αν παίρνουμε χρήματα από το Horizon 2020 που βασίζεται σε χρήματα που σε επιχορηγήσεις, αυτό θα κάνουμε και εδώ. Αν θέλετε να αυξήσει η μόχλευση και να προσελκύσετε ιδιωτικού επενδυτές, πώς θα το κάνετε χωρίς να βάζετε το δημόσιο να παίρνει τον κίνδυνο και τους ιδιώτες να ε, κερδίζουν μόνο. Μέχρι τώρα δεν έχουμε δει καμία βελτίωση σε αυτό. Οπότε θα ήθελα να μας εξηγήσετε καλύτερα πώς θα γίνει η σύνδεση αυτή μεταξύ του δημοσίου και του ιδιωτικού. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Βάλλη έχει τώρα το λόγο εκ μέρους Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων. Ναι. Ε, νόμιζα ότι είχαμε μία χρονοθυρίδα να ομάδα, αλλά τέλος πάντων. Ε, η δική μου ερώτηση αφορά και απευθύνεται στον Διευθυντή του Οργανισμού Περιβάλλοντος. Ήθελα να μου πείτε τη γνώμη έχετε για τα έργα που έχουν υποβάλει τα κράτη-μέλη για την αποθήκευση άνθρακα και τι έγινε με τα ανάλογα προγράμματα της Ισπανίας, πώς ε, αποδείχθηκε η περιβαλλοντική βιωσιμότητα. Ε, είδαμε ότι με τέτοιου είδους συγκεκριμένα έργα υπάρχει τελικά αποσταθεροποίηση του, υποδα... του υπεδάφους. Το περιβάλλον ε, ουσιαστικά πλήττεται και υπάρχουν μετασυσμοί και ούτω καθεξής. Αυτό μας ανησυχεί πολύ. Υπάρχει ιδιαίτερη πίεση από τις ανάλογες ομάδες για τέτοια έργα και πολλά εμφανίζονται μεταξύ των υποψηφιότητων. Τι γνώμη έχετε λοιπόν για τέτοιου είδους έργα. Ευχαριστώ. Πρόεδρος, και τώρα ολοκληρώνουμε με τους δύο εισηγητές ε, της Επιτροπής Ήτρε, των Επιτροπών Ήτρε και Τραν, η κυρία Φαν Μπρέντ πρώτη από την Επιτροπή um, Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε και ευχαριστώ πολύ όλους τους ομιλητές μας. Θέλω να ρωτήσω κι εγώ κάτι, αλλά θέλω μια συγκεκριμένη απάντηση, γιατί είμαι κι εγώ, όπως και άλλοι, υπεύθυνοι για τη γνωμοδότηση, με αρμοδιότητα μόνο να δούμε από πού θα έρθουν τα χρήματα. Από το Horizon 2020. Οι ομιλητές βέβαια σωστά λένε ότι δεν μπορεί να βγάλουμε τα χρήματα από τον προπολογισμό για τις υποδομές ή για την έρευνα τη στιγμή που τόσο ισορροπημένα τα έχουμε προβλέψει για να τα βάλουμε στην εγγύηση. Πρέπει να βρούμε εναλλακτικέ λύσει. Η ερώτησή μου όμω, πιο συγκεκριμένα έχει με το είδο των έργων και ο κύριο Μάιστατ σε ένα βαθμό έχει απαντήσει γιατί έχει βέβαια εμπειρία από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και αυτό που είπε και ο κύριο Μπράινιξ. Θέλω να πω ότι συμφωνώ μαζί του 100%. Αλλά ακριβώ για να υπάρξει αυτό το πιο συγκεκριμένο στον κανονισμό δεν έχουμε αρκετά. Η ερώτησή μου λοιπόν είναι απλή, αλλά βέβαια η απάντηση δεν είναι απλή. Πώς θα φροντίσουμε στο άρθρο 5, παράγραφος 2, εκεί που είναι τα διάφορα μέρη, θα συμπεριλάβουμε τα σωστά διότι δεν είναι κλειστός αυτός ο κατάλογος. Μπορεί να καταλήξουμε να βάλουμε και μία μονάδα επεξεργασίας άνθρακα. Οπότε πώς θα φροντίσετε στο σημείο 5.2 τα έργα θα καθορίζονται έτσι που η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων θα πηγαίνει προς τη σωστή κατεύθυνση και μόνο. Ευχαριστούμε. Η κυρία Γιάλα Σέντερ τώρα. Ευχαριστώ. Θέλω να ρωτήσω, δεν ξέρω ποιον ακριβώς, ίσως και τον κύριο Μάιστατ, σε σχέση με την συμπληρωματικότητα. Λείπουν διάφορα εκατομμύρια και λέμε ότι ίσως κάθε χρόνο να τα βρίσκουμε για να καλύπτεται το Ταμείο. Κύριε Ολάντ, είπατε ότι τα δάνεια από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων δεν θα υπολογίζονται στο, στην αξιολόγηση της δημοσιονομικής προσαρμογής. Σωστά σας κατάλαβα. Εγώ νομίζω ότι ήταν το αντίθετο. Αλλά αν είναι έτσι, πώς Συγκεκριμένα λοιπόν θα λάβουμε υπόψη μας τα κίνητρα για τις δημόσιες επενδύσεις, για τις μεταφορές. Γιατί όπως τα ακούσαμε, για τις μεταφορές συνήθως για αυτοκινητοδρόμους είναι. Και εσά τώρα, κύριε Μέστε, θέλω να σας ρωτήσω επίσης κάτι. Συμφωνώ μαζί σας. Είναι, ναι, σωστό, Silicon Valley, ναι. Αλλά του περιβάλλοντος εννοώ. Όμως, η απασχόληση που δημιουργείται. Μόλις και με τα τη βλέπουμε. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν μας δίνει νούμερα, μας λέει ότι υπάρχει, αλλά δεν είναι ορατές αυτές οι θέσεις απασχόλησης για τους πολίτες. Γι' αυτή λοιπόν την κυκλική οικονομία πρέπει να ξέρουμε ότι δεν βλέπουμε τα νούμερα έτσι ώστε να αποφύγουμε την μεταφορά επιχειρήσεων ή τις απότομες αναδιαρθρώσεις των επιχειρήσεων. Ίσως εσείς μπορείτε να μας βοηθήσετε. Στον κύριο Μπάρτη θέλω να πω, μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Έρχεστε από το οικό, ναι. Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων λοιπόν, πιστεύετε ότι έχει τη δυνατότητα να καλύψει τις πραγματικές ανάγκες των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, του Νότου, τις μικρές, των ε, ελευθερών επαγγελματιών και κάτι για τον κύριο Μαϊστέτ. Πώς να αποφύγουμε τη προσωρινή εξαίρεση προκειμένου να βοηθήσει να αποφεληθούν αυτοί που έχουν μεγαλύτερο έλλειμμα από 3% αυτές τις χώρες. Πρόεδρος, πολλές σημαντικές ερωτήσεις, αλλά μόνο δύο λεπτά έχει ο κάθε ομιλητής μας για να δώσει απαντήσεις. Ο κύριος Μέιστατ πρώτα. Ευχαριστώ Πρόεδρε, δύσκολο με τόσο λίγο χρόνο να απαντήσω πλήρως σε όλες αυτές τις τόσο εύστοχες ερωτήσεις που τέθηκαν. Πολλές ερωτήσεις αφορούν το Ταμείο των Εγγυήσεων. Άρθρο 8 του σχεδίου κανονισμού. Εκεί προβλέπεται ότι ο στόχος είναι στο ταμείο αυτό να έχουμε 50% του συνόλου των εγγυήσεων που θα προβλέψει η Ένωση. Ένα ποσό που είναι αρκετά ε, ασφαλές αλλά θα δικαιολογηθεί μόνο αν η ΕΤΕ αναλάβει πολύ περισσότερους κινδύνου από ό,τι τώρα. Για να σας δώσω ένα μέτρο σύγκριση για τα ταμείο Εγγύησεων για τις εξωτερικές δράσεις της ΕΤΕ, δράσεις εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης και ε, κυρίως της χώρας ΑΚΕ, όπου οι κίνδυνοι είναι αρκετά συχνά υψηλοί, το ταμείο εκεί, οι εγγύησει, ε, χρηματοδοτούνται κατά 9% από τις δεσμεύσεις της ΕΤΕ. Εδώ τα πράγματα είναι κάπω ε, διαφορετικά, διότι λέμε 9% του συνόλου των δεσμεύσεων. Τώρα λέμε ότι πρέπει στο Ταμείο να ε, βάλουμε το 50% του συνόλου των εγγύησεων που παρέχονται. Θα δικαιολογείται κάτι τέτοιο εάν όντω η ΕΤΕ αναλάβει πολύ περισσότερο κίνδυνο. Και αν υπάρχει μια πιθανότητα στις δύο να ε, κινητοποιηθεί αυτή η εγγύηση. Όμως θα πρέπει να γίνει αυτό προοδευτικά. Δηλαδή στα 50% πρέπει να φτάσουμε ενώ η ΕΤΕ απευθύνεται στο και χρησιμοποιεί το Ευρωπαϊκό Στατικό Ταμείο. Δηλαδή, καθώς υπάρχουν δάνεια από την ΕΤΕ. Ιδάλλως, το 50% των 16 δις δεν χρειάζεται να το καταρτήσουμε φέτος. Η ΕΤΕ μπορεί να χρειαστεί μόνο 16, να μην χρειαστεί 16 δις ε, φέτος, αμέσως. Θα πρέπει λοιπόν σταδιακά από την ΕΤΕΝ να δημιουργηθεί αυτό το Ταμείο Εγγύσεων. Αυτό ήθελα να το επισημάνω. Και επίσης πώς θα τροφοδοτείται αυτό το Ταμείο Εγγύσεων, πού θα βρούμε αυτό το 50%. Είναι προφανώς το πιο δύσκολο ερώτημα. Και μιλώ εδώ τελείως άνετα και ελεύθερα. Εγείρει ερωτήματα. Γιατί διότι από τη μια θα πάρουμε κονδύλια από το Connecting Europe Facility και από την άλλη από το Horizon 2020. Αυτό ρώτησε και η κυρία Φαν και είναι πολύ εύστοχη ερώτηση. Ποια είναι η συλλογιστική της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που είναι και πολύ συγκεκριμένη. Λέει ότι Αντί να χρησιμοποιήσουμε αυτά τα δημοσιονομικά μέσα ως ευγρογήσεις, ας τις βάλουμε στο εύση, οπότε η μόχλευση θα λειτουργήσει. Η μόχλευση δεν θα είναι πάντοτε αναγκαστικά 1 προς 15, αλλά μπορεί να είμαστε στο 1 προς 10. Και πάλι, αντί να δώσουμε 100 ως επιχορήγηση, μπορούμε να χρηματοδοτήσουμε πολύ περισσότερο μέσω του εύση, μέσω της μόχλευσης, με 1000, μπορεί και 1500. Βλέπουμε τη συλλογιστική, όμως ε, προκύπτουν άλλα ερωτηματικά εδώ. Πολύ γρήγορα σας παρακαλώ. Δεν θα θίξω τα υπόλοιπα ερωτήματα. Όμως νομίζω ότι είναι ένα από τα πιο σημαντικά σημεία της όλης συζήτησης. Δηλαδή, δεν θα είναι πάντοτε οι ίδιοι δικαιούχοι. Όπως στην έρευνα στο Horizon 2020 είναι σαφέ ότι η ΕΤΕ έχει σχετική πείρα, ιδίω με, ε, με το μηχανισμό ε, κατανομής του κινδύνου. Εκεί η εμπειρία τη έχει διδραματίσει ρόλο μόχλευση. Όμω, ασχολήθηκε με εφηρμοσμένη έρευνα, με έρευνα που γρήγορα θα οδηγούσε σε εμπορική πραγματική επιστροφή και κέρδο. Έτσι μπορούσε ο ιδιωτικό τομέα να περάσει σε χρηματοδότηση τέτοιου είδου έρευνα. Αυτό έχει γίνει ω τώρα. Κινδυνεύουμε να έχουμε λιγότερα μέσα για να χρηματοδοτήσουμε την έρευνα, τη βασική έρευνα, την θεωρητική. Και αυτό εξηγεί τι αντιδράσει τη επιστημονική κοινότητα. Είναι ένα θέμα που πρέπει να μα απασχολήσει. Ένα άλλο θέμα είναι το Connecting Europe Facility. Εδώ δεν θέλω να προδικάσω τι θα πούνε οι εμπειρογνώμονε των μεταφορών, όμω κάποιε επενδύσει στον τομέα των μεταφορών έχουμε οπωσδήποτε ανάγκη από άμεσες επιδοτήσεις. Δεν μπορούμε να τις ε, χρηματοδοτούμε μόνο με αυτό το θέμα, με την διάσταση της μόχλευσης και τον ιδιωτικό τομέα. Οπότε πρέπει να δούμε αν θα υπάρχουν αρκετές δυνατότητες για κάποια από τα προγράμματα που όλοι αναγνωρίζουν ότι είναι προτεραιότητας, ιδίως στον τομέα των μεταφορών, των σιδηροδρομικών μεταφορών. Εκεί πρέπει να δούμε αν υπάρχει ακόμη η δυνατότητα να δοθούν επιδοτήσεις. Πρόεδρο, ευχαριστούμε, ευχαριστούμε πολύ. Ο κύριος Γκρούνιξ. Ευχαριστώ, Κατά πρώτον, να απευθυνθώ να, μιλήσω για το θέμα του επεδάφους και της αποθήκευσης άνθρακα. Γνωρίζοντας το τι έχουμε εμείς στα χέρια μας ως Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος, δεν έχουμε σοβαρές μελέτες για το θέμα αυτό. Προτιμώ λοιπόν να πω ότι προς στιγμήν είμαστε εν αγνία για αυτό το θέμα. Αλλά για τα επιμέρους έργα που αναφέρατε δεν έχω συγκεκριμένη γνώση. Υπάρχουν πάντω σχετικέ διαδικασίε στην Ευρώπη και αρχέ που ε, καθορίζουν τη χάραξη πολιτική και ε, ενσωματώνονται στην ε, συνθήκη τη Λισαβόνα όπω η αρχή τη προφύλαξη ή η χρήση του προδοπαροντικού αντικτύπου και τη μελέτη του. Αργότερα μέσα στη χρονιά θα διοργανώσουμε σε συνεργασία με την επιστημονική κοινότητα ένα σεμινάριο που τον ονομάσαμε οι ανταγωνιστικές αξιώσεις του υπεδάφους και εκεί θα επικεντρωθούμε στον κανονισμό, στους διάφορους κανόνες που έχουμε για το υπέδαφος. Ως προς το πώς θα βεβαιωθούμε ότι το άρθρο 5.2 και ερωτήθηκε αυτό από τον κύριο Κάρα, αν καλά κατάλαβα, πώ θα μα οδηγήσει αυτό στα προσδοκόμενα αποτελέσματα. Ω οργανισμό συγκέντρωση γνώσεων, θα ήθελα να επικεντρωθώ στα δύο παραδείγματά σα. Όταν μιλήσατε για ένα εργοστάσιο παραγωγής ενέργειας που ε, κινείται με άνθρακα. Εάν δούμε με σοβαρότητα την προοπτική του 2050, το ερώτημα είναι, θέλουμε να επενδύσουμε στο να ε, γίνει το σημερινό σύστημα που βασίζεται στον άνθρακα πιο αποδοτικό, πιο αποτελεσματικό, γνωρίζοντας τα όρια του, ή θέλουμε να επενδύσουμε στη μετάβαση προς ένα νέο είδο παραγωγή ενέργεια, ένα νέο σύστημα παραγωγής ενέργειας. Αυτό είναι ένα από τα κριτήρια που θα πρέπει να μας καθοδηγούν και σε ό,τι αφορά το παράδειγμά σας για την κινητικότητα, από το 1990 ο τομέας των μεταφορών έχει προσθέσει 20% εκπομπές στο σύνολο. Είναι ο μόνος τομέας που έχει ε, διεγκωθεί στην Ευρωπαϊκή. το 2050 ο τομέας κινητικότητα και μεταφορών στην Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να μειώσει τις εκπομπές του κατά 60%. Πώς λοιπόν θα επενδύσουμε στην αποδοτικότητα και στο σύστημα κινητικότητας όπως ισχύει σήμερα. Αυτό θα κάνουμε, θα το βελτιώσουμε απλώς ή θα κοιτάξουμε να επενδύσουμε στο μέλλον που να δημιουργήσει ένα δίκτυο μεταφορών χαμηλής κατανάλωσης άνθρακα. Αυτό είναι η πραγματική προτεραιότητα και εκεί θα χρειαστεί πραγματική καινοτομία. Και πολύ σύντομα, σε ό,τι αφορά τι ερωτήσει για τι νέε θέσει εργασία και την περισσότερη τη νέα απασχόληση. Αν είναι εντελώ καινούρια και πώ σχετίζονται με την βίαιη, όπω είπατε, αναδιάρθρωση τη οικονομία σε κάποιε περιοχέ. Σε ό,τι αφορά την μακροοικονομική διάσταση και ε, την κοινωνική ταυτόχρονα αυτού του είδους επενδύσεων, ε, που ήταν ένα από τα βασικά στοιχεία της ακρόασης και της ε, όλης συζήτησης, νομίζω ότι πρέπει πάντοτε να κοιτάμε τον καθαρό αντίκτυπο και γνωρίζουμε όλοι από τα αποδεκτικά στοιχεία ότι ο καθαρός αντίκτυπος της κατεύθυνση που υπέδειξα ήταν θετικός. Δεν σημαίνει ότι κάθε, ένα, κάθε μια εταιρεία, κάθε επιχείρηση, ο καθένας μεμονωμένα θα επωφεληθούν από αυτή την άγουσα. Αλλά αν κοιτάξουμε πολλές πόλεις στην Ευρώπη όπου ακόμη κάποιοι δρόμοι έχουν τα ονόματα των ε, όσων κατασκευάζαν τα αμάξια που έσωναν τα άλογα. Θα δούμε πώς ε, η βιομηχανία αυτή βοήθησε την Ευρώπη να αναπτυχθεί. Εδώ λοιπόν έχουμε όχι την αντίφαση και την αντίθεση ανάπτυξης και καταστροφής, αλλά το κατά πόσον αυτή η κοινωνία θα επικεντρωθεί σε νέα ανάπτυξη, σε νέες θέσεις εργασίας, με νέες συνέπειες που από κοινωνική άποψη σίγουρα θα έχουν κάποιες επιπτώσεις, όμως η Ευρώπη έχει την ιστορία και τις γνώσεις για να τα αντιμετωπίσει αυτά με τρόπο σοβαρό. Ευχαριστώ. Θα δώσω την Προεδρία στον κύριο Αρτουή από την Επιτροπή Προπολογισμών. Ευχαριστώ, Ρομπέρτο. Ολοκληρώσαμε, συνεπώς, με το πρώτο τμήμα. Τώρα παρακαλώ να έρθουν στο βήμα ή όχι. Όχι. Α, συνεχίζουμε. Α, ο κύριος Σαμπάντ τότε. Παρακαλώ, έχετε το λόγο κύριε Αμπάτ. πέντε πράγματα. Πολλά έχουν ήδη υποθεί. Το πρώτο που θέλω να πω είναι να τονίσω ότι το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων είναι ένας πυλώνας μόνο. Μην επικεντρωνόμαστε μόνο σε αυτόν, γιατί δεν είναι το πιο σημαντικό. Ας δούμε όλο το πρόγραμμα, γιατί και άλλοι δύο πυλώνες είναι πολύ σημαντικοί. Το δεύτερο έχει να κάνει με την μόχλευση. Το ρωτήσατε πολύ. Φυσικά και μιλάμε για μια μόχλευση 15 από τις επενδύσεις του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων μέχρι το τελικό σύνολο. Εντάξει, είναι δύσκολο, αλλά με τις επενδύσεις του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων θα φτάσει στα 63 δισεκατομμύρια επενδύσεις με τη μόχλευση. Επιτρία για την ίδια την ΕΤΕ. Τώρα οι επενδύσεις θα προσελκύσουν ιδιωτικές επενδύσεις με πολλαπλασιαστή 5. 3 επί 5, 15. Τρίτον, η δημιουργία του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων ακολουθεί τις πρακτικές που έχουμε και σε άλλες χώρες. Το είπα και στην αρχή. Και στις Ηνωμένε Πολιτείε γίνεται αυτό. Υπάρχουν χώρες που έχουν αγορές με πολύ πιο μακροχρόνιες επενδύσεις. Τέταρτον, είναι αλήθεια. Το ότι ένα έργο δεν έχει σχέση με την αρχική ιδέα δεν έχει να κάνει με την μόχλευση. Και το τελευταίο έχει να κάνει με τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και θα συνεχίσω ισπανικά, λέει ο μιλητής. Πράγματι υπάρχουν διάφορες χώρες, Ισπανία μεταξύ άλλων, που έχει πιο μικρές επιχειρήσεις. Η μέση μικρομεσαία επιχείρηση στη Γερμανία είναι πιο μεγάλη από την αντίστοιχη Ισπανική. Όντως, χάνονται πολύ περισσότερες μικρομεσαίες επιχειρήσεις, είναι αλήθεια αυτό στην Ισπανία. Οι εγγύησει. Γι' αυτό ακριβώς είναι πολύ πιο χρήσιμες στις χώρες εκείνες που έχουν πιο μικρές μικρομεσαίες επιχειρήσεις, γιατί ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος για τις τράπεζες που τις δανείζουν. Βάσει της Βασιλείας 3, αν ένα μεγάλο μέρος της πελατεία σου είναι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ο κίνδυνος αυξάνει, άρα το κόστος για την τράπεζα είναι μεγαλύτερο. Εξού και οι εγγύησει έχουν μεγάλο βάρος για αυτή την περίπτωση. Πάντως, το σκέλος που χρηματοδοτεί το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων. Υπάρχουν εγγύησει, είπαμε, αυτό είναι το ένα, και το άλλο είναι η, τα ιδιωτικά κεφάλαια, τα κεφάλαια κινδύνου. Σαν εναλλακτική μορφή χρηματοδότησης, και στην Ισπανία αλλά και σε άλλες οικονομίες. Είναι μια ευκαιρία δηλαδή, αυτή είναι η απάντησή μου, ιδιαίτερα για τις χώρες που έχουν πιο μικρές επιχειρήσεις όπως είναι η Ισπανία. Πρόεδρος, ευχαριστούμε κύριε Παντό. Κύριος Χόλαντ τώρα. Τρία ε, θέματα έχω να σας πω. Πρώτο, Φάβιο Ντεμάζη και εσείς. Πώς δηλαδή ο δανεισμός από την ΕΤΕ δεν λογαριάζεται στο δημόσιο χρέος και πώς μπορούν τα ταμεία αυτά να βγουν έξω από τα κριτήρια Μάστριχτ. Μα διότι δεν είναι χρήματα των ε, κρατών μελών. Δεν είναι εθνικό χρέος. Δεν συνυπολογίζεται λοιπόν στο δημόσιο χρέος, διότι αν συνυπολογιζόταν τότε θα ήταν διπλό παθητικό. Αυτό είναι η υπόθεση της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Δεν είναι παθητικό των χωρών στις οποίες δανείζει. Δεν είχα ξεκαθαρίσει τόσο πολύ κάτι το Δεκέμβρη. Σύμβουλοι επιτρόπων δεν γνώριζαν, σύμβουλοι επιτρόπων δεν γνώριζαν ότι ο δανεισμός από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων δεν συνυπολογίζεται στο δημόσιο χρέος. Ο κύριος Σόιπλε, ο οποίος έχει μανία με, με, με το χρέος και το σούλτ βέβαια που σημαίνει και χρέος αλλά και φταίξιμο ενώ βέβαια η άλλη λέξη η πίστη, η πίστοση προέρχεται από το λατινικό credo, credit, πιστεύω δηλαδή σε σένα. Έτσι λοιπόν από εκεί μέσα βγαίνει όλη αυτή η διάσταση. Και τώρα πιο σύντομα. Δεν χρειάζεστε επένδυση σε κίνδυνο γιατί να ασχοληθείτε με τέτοια πράγματα τα οποία σε επιδοτήσει του δημοσίου ένα από τα ισχυρά σημεία του Ζακ Τελόρ και εγώ τον συμβούλευα τότε ήταν ότι πίστευε ότι πρέπει να υλοποιήσει την ενιαία ευρωπαϊκή πράξη για την ενιαία αγορά και για την ευρωπαϊκή συνοχή και η ανάκαμψη πρέπει να είναι βασισμένη σε κοινωνική επένδυση δηλαδή σε παιδεία, υγεία, αστική ανακαίνιση. Υπάρχουν ανάγκες σε όλα αυτά και θα δημιουργήσουν και ζήτηση στον ιδιωτικό τομέα. Χτίζει ένα νοσοκομείο, αυξάνονται και οι ανάγκες για φάρμακα, λειτουργεί. Τέλος, σε σχέση Καθρίν Βαν Μπρέμπτ, σας παρακαλώ για την έκθεσή σας. Μην θέτετε απλώς ερωτήσεις. Μην εκφράζετε μόνο αμφιβολίες. Ξεκινήστε από ένα βασικό, ότι μέσα στην πρόταση δεν, υπάρχουν, δεν υπάρχει πραγματικό χρήμα. Ενώ σε κοινή χρηματοδότηση από Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων μπορούν να υπάρξουν. Τα κριτήρια του ειδικού προγράμματος δράσεως του Άμστερνταμ πράσινες τεχνολογίες, μικρές μεσαίες επιχειρήσεις, υγεία, παιδεία, είναι ήδη αρκετό. Τελευταίο, μετά από το ειδικό πρόγραμμα δράσεως του Αμστερνταμ, το οποίο μάλιστα το είχε προτείνει τότε ο Αντώνιο Κουτιέρες και το καλωσόρισε η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, τετραπλασίασε τις επενδύσεις της η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων μεταξύ 1997 και 2007. Με τη βοήθεια των προγραμμάτων αυτών που συνέβαλαν στην συνοχή. Υπάρχουν λοιπόν τα απαραίτητα εργαλεία. Δεν χρειάζεται να επινοήσετε άλλα. Μην συνεχίσετε να θέτετε ερωτήσεις για το ταμείο αυτό, το EFSI δηλαδή, το οποίο δεν πρόκειται να επιτύχει. Έχει προφυλακτικό χαρακτήρα, ναι, αλλά στην πραγματικότητα παρεμποδίζει την περαιτέρω συζήτηση βασιστείτε στα εργαλεία που είχε σχεδιάσει και υλοποιήσει τότε ο Ντελόρ πριν από 20 χρόνια. Ευχαριστώ τους τέσσερις ομιλητές μας που μας έδωσαν τις απαντήσεις τους. Ε, μοιράστηκαν μαζί μας τις απόψεις τους. Να ευχαριστήσω τον κύριο Μέστατ, τον κύριο Αμπάντ, τον κύριο Ολόντ, και να προσκαλέσω τώρα τους ομιλητές αυτού του δεύτερου τμήματος της ε, ακροασής μας, τον κύριο Κέλλερ και τον κύριο Γκρός, να έρθουν εδώ για να μας ε, απευθυνθούν. Το δεύτερο αυτό μέρος της ακρόασης αφορά τις πρακτικές εφαρμογές και την ιδιωτική, τις ιδιωτικές επενδύσεις. Να δώσω το λόγο για 10 λεπτά στον κύριο Κέλλερ, πρόεδρε του Ιδρύματος Κένουπ. Κύριε Κέλλερ, έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ που μας δίνατε την ευκαιρία να σας απευθυνθούμε. Η κοινότητα των ιδιωτικών επενδύσεων σε καμία περίπτωση δεν έχει πρόβλημα ρευστότητας και έχει και πολύ μεγάλη όρεξη για μια σταθερή Ευρώπη. Αυτό τείνουμε να το ξεχνάμε. δυστυχώς πολλές από τις επενδυτικέ ευκαιρίες έχουν να κάνουν με τις λειτουργίες της αγοράς και των αγορών όπου δεν υπάρχουν αρκετά κίνητρα και υπάρχουν παροχημένοι κανόνες. Για να απελευθερωθεί η δυνατότητα του ιδιωτικού τομέα στις επενδύσεις χρειάζεται μια συγκεκριμένη πλατφόρμα με επενδυτές για την έρευνα και ανάπτυξη, τους ρυθμιστές και κάτι που δεν έχω ακούσει ακόμα τώρα σήμερα, την κοινωνία των πολιτών. Επιτρέψτε μου να πάω λίγο πιο γρήγορα με μια επιτάχυνση και να σας παρουσιάσω το Ίδρυμά μας, το Κένουπ, που είναι από αυτές τις πλατφόρμες που ήδη κάνει πολλά από αυτά που προτείνει το πρόγραμμα Juncker ή που ελπίζει να κάνει, προσδοκά το πρόγραμμα Juncker. Επόμενη διαφάνεια. Τι έχουμε κάνει ως τώρα. Έχουμε εντοπίσει πολύ συγκεκριμένες ευκαιρίες στην αγορά των επενδύσεων ε, όπως αναδύονται λόγω των δημογραφικών εξελίξεων. Οι δημογραφικές εξελίξεις έχουν επιπτώσει στην υγεία και τη σχετική αγορά και πολύ συγκεκριμένα στις ευκαιρίες επενδύσεων που τώρα ε, ε, αξιοποιούν στην Κίνα και τις Πολιτείες αλλά δυστυχώς όχι ακόμα στην Ευρώπη. Σε, μια διετή, σε ένα διετή ορίζοντα, και αυτό είναι ακόμη μέρος του προγράμματος Juncker, έχουμε μιλήσει με consultant, με συμβούλους από τον τομέα των τραπεζών των επιχειρήσεων και με πολλά επιστημονικά ιδρύματα, εντοπίζοντα 26 περιπτώσει ευκαιριών όπου θα μπορούσε η Ευρώπη να αναλάβει πρωταγωνιστικό ρόλο στην ε, διεθνή αγορά. Όχι λοιπόν να προλάβουμε απλώ τι εξελίξει, αλλά να έχουμε ηγετικό ρόλο. Οι ε, περιπτώσει αυτέ είναι τα εμβόλια για του ενηλίκου, ε, Ένα τομέα βιομηχανία όπου έχει πρωταγωνιστικό ρόλο η Ευρώπη, είχε μάλλον επί πολλά χρόνια και τώρα έχει χάσει την πρωτιά τη. Τα ε, καινοτόμα εμβόλια, όχι μόνο για την ογκολογία και άλλου τομεί, την υψηλή ποιότητα υγειονομική περίθαλψη με προστιθέμενη αξία για του ασθενεί, τι ανεξάρτητε λύσει καθώ και την, ε, την, τον εξυγχρονισμό της ε, περίθαλψης. Αυτό το σύνολο ε, βιομηχανικών, ε, επιχειρησιακών μάλλον επιλογών θα δείξει εάν μπορούμε να αναλάβουμε πρωταγωνιστικό ρόλο διεθνώς από την Ευρώπη ή όχι και κατά το μοντέλο μας είναι ε, σκόπιμο. Τώρα, γιατί ακόμη δεν τα έχουμε καταφέρει. Είναι απλό να το κατανοήσει κανείς. Έχουμε ένα σύστημα κινήτρων που είναι ελάχιστο ομογενοποιημένο ιδίω για αυτού του τομεί. Δηλαδή μιλάμε για έναν χώρο του κόσμου που ευφυεί άνθρωποι σε εξαιρετικούς οργανισμούς συστηματικώς λαμβάνουν ηλίθιε αποφάσεις. Αυτό είναι σαφές. Η προπόθεση για τις επενδύσεις ε, καταργείται κατά αυτόν τον τρόπο. Οπότε ε, έχουμε περιέλθει σε μια κατάσταση όπου οι επιχειρήσεις, η ε, κλάδοι αυτή δραστηριότητας ε, επιδοτούνται ιδιαίτερως παγκοσμίω. Όμως στην Ευρώπη έχουμε ελάχιστε νεοφυεί επιχειρήσει, ελάχιστε μικρομεσαίε, μικρομεσαίες πρωτοβουλίες που θα μπορούσαν να είναι μελλοντικές Microsoft, Intel, Facebook ή οτιδήποτε ανάλογα. Και Πολύ απλά, αν κοιτάξουμε αυτούς τους βιομηχανικούς κλάδους, δεν υπάρχουν εταιρείες που να ε, επιθυμούν τον πρωταγωνιστικό ρόλο στην Ευρώπη. Επόμενη διαφάνεια. Έχουμε λοιπόν μια σύμπραξη εδώ ε, πολλών τομέων για το μέλλον και πρέπει να πούμε ελάτε όλοι μαζί με μια κοινή προσπάθεια σε ανθρώπους που δεν κάθονται γύρω από το ίδιο τραπέζι. Ελάτε να εκμεταλλευτούμε αυτή την ευκαιρία. Πρέπει τα κράτη-μέλη να αναλάβουν κάποια πρωτοβουλία. Η δημοκρατία της Μάλτας και η δημοκρατία της Κροατίας με στήριξη από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας πρέπει να πούν ότι μπορούμε να αναλάβουμε ευθύνη στον εξυγχρονισμό μας στο επίπεδο του κράτους μέλους κατά πρώτον με την συμμόρφωση με τους διάφορους κανονισμούς που προβλέπονται. Και σε αυτούς τους έξι τομείς μπορούμε να φέρουμε σε συνεργασία τους πιο ενδιαφέροντες φορείς από όλο τον κόσμο για να εξυγχρονίσουμε το σύστημα καινοτομίας και να δημιουργήσουμε έναν διάβλο για την πρόθεση των έργων. Όλα αυτά θα πετύχουν μόνο αν συμμετέχει η κοινωνία των πολιτών. Εσείς ε, σχεδιάζετε τους νόμους, αλλά θα τους σχεδιάσετε σωστά μόνο εάν συγκεκριμένα τμήματα τα της κοινωνίας των πολιτών σας δώσουν τη συνεισφορά τους και τη στήριξή τους. Πολύ το επενδυτικό περιβάλλον είναι πολύ ανασφαλές. Αν σκεφτούμε την, την παρατήτηδα και τα εμβόλια τη, η όλη συζήτηση για την κοινωνία των πολιτών έχει να κάνει με τι απειλέ για τη δημόσια υγεία, αλλά και την, την απώλεια, την έλλειψη μάλλον επενδύσεων σε αυτό το τομέα. Έχουμε λοιπόν ένα σύστημα που είναι αρκετά απλό και συνολικά στοχεύει στις σχετικά μικρές στοχεύει στις μικρές ιδιωτικές επενδύσεις και σε ένα σημαντικό παράγοντα μόχλευσης που έχει να κάνει με την αποδέσμευση των ιδιωτικών επενδύσεων αλλά και την αξιοποίηση των ε, σχέσεων συνεργασίας με άλλα υπάρχοντα προγράμματα του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα όπου υπάρχουν. Κυρίως ο σκοπός είναι να διαρθωθούν όλα αυτά σε ένα μικρό ταμείο, ένα μικρό χώρο ε, που θα λειτουργήσει σε μια επιχείρηση που δεν χρειάζεται ιδιαίτερη χρηματοδότηση μια επιχείρηση συνήθως χρειάζεται για να λειτουργήσει ένα δάνειο όπως ε, το έχετε ορίσει εσείς με, μια, ένα πρόγραμμα αποπληρωμής ε, και θα πρέπει διαρκώς να υπάρχει επένδυση στη συγκεκριμένο τομέα καινοτομία στην Ευρώπη. Επόμενη διαφάνεια. Τι πραγματικά χρειαζόμαστε. Τρία πράγματα. Μια διαδικασία λήψης αποφάσεων για το Ταμείο που είναι τελείω ανεξάρτητη από τα συμφέροντα των ενδιαφερομένων, δηλαδή τα αρχικά συμφέροντα των ιδρυτών, την ίδια, τον ίδιο το βιομηχανικό κλάδο της επιχειρήσης και ε, πιο συγκεκριμένους ε, ενδιαφερομένους. Δεύτερο στοιχείο που χρειαζόμαστε είναι να είμαστε σε θέση να διαχειριστούμε το Ταμείο σαν να είναι ε, ε, μια οντότητα που θα παράγει κέρδος με την κατάλληλη μόχλευση και έπειτα εκφύσεως τα διάφορα εργαλεία του συστήματός μας καλύπτονται από τα περισσότερα κράτη-μέλη τις 22 χώρες που συμμετέχουν στο σύστημά μας κάτι που δεν αφορά μόνο τα μικρά ή τα μεγάλα κράτη αλλά την, ούτε την ανακατονομή των κονδυλίων απλώς την δημιουργία αξίας για την Ευρώπη την χρήση των ε, ε, ε, λιγοστών δημοσίων κονδυλίων για την απελευθέρωση ιδιωτικών κεφαλαίων που αυτή τη στιγμή τα επενδύουν αλλού. Γι' αυτό η πλατφόρμα για τις επενδύσεις είναι σκόπιμη και πραγματικά θα συνιστούσαμε στο Κοινοβούλιο να σκεφτεί ότι ό,τι κάνει, ό,τι αποφασίζει θα πρέπει να είναι πάρα πολύ συνετό για τις επιχειρήσεις, για τις ενδράσεις που θα προβλέψει και για το τι μπορεί να ε, γίνει. Ευχαριστώ για το χρόνο σας. Merci. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Κέλλερ. Το λόγο έχει τώρα ο κύριος Ματιέ Γκρός, ο οποίος είναι εμπειρογνώμων στον ιδιωτικό τομέα και που όρισε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συντονιστή διευρωπαϊκών δικτύων μεταφορών. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Δεν είμαι από τον ιδιωτικό τομέα. Ε, και 20 χρόνια στο δημόσιο πιο πολύ είμαι. Ασχολήθηκα βέβαια με τα διευρωπαϊκά δίκτυα όλο αυτό τον καιρό. Λοιπόν, σήμερα θα σας πω πώς ένα ταμείο που ήδη υπάρχει, πώς λειτουργεί, ποιες είναι οι προκλήσεις που αντιμετωπίσαμε σε αυτό και ποιες είναι οι προοπτικές για το μέλλον στα πλαίσια της διευκόλυνσης συνδέοντας την Ευρώπη. Οι προκλήσεις μας, θα τις επαναλάβω σύντομα. Έχουμε όλο και περισσότερο ζήτηση μεταφορών και από την άλλη μεριά έχουμε και την εξέλιξη που γνωρίζουμε με το διοξίδιο του άνθρακα. Οι μεταφορές είναι ο μόνος τομέας, ακόμα και αν το συγκρίνουμε με τη βιομηχανία, όπου έχει αυξηθεί το διοξίδιο του άνθρακα και έχουμε θέσει ένα σαφή στόχο για το 2020. Η δεύτερη πρόκληση είναι να δούμε την εξέλιξη της ζήτησης που εκτιμούμε ότι θα είναι 50% για τις επιβατικές μεταφορές και 80% για τις μεταφορές εμπορίων και να το συγκρίνουμε αυτό με την έλλειψη επενδύσεων στις υποδομές. Βλέπετε εδώ την εξέλιξη. Συγκρίνουμε τι γίνεται επίσης στις ΗΠΑ και στην Ευρώπη όσον αφορά τις επενδύσεις. Και αύριο εδώ στις Βρυξέλλες να ξέρετε ότι θα παρουσιαστεί και μία μελέτη για τις σιδηροδρομικές μεταφορές και την εξέλιξή τους. Και αυτό μπορώ να σας πω ήδη από τώρα είναι ότι σε χώρες ακόμα και όπως η Γερμανία έχουμε λιγότερες επενδύσεις κατά 300 εκατομμύρια, στη Γαλλία 400 εκατομμύρια, λιγότερες από αυτό που θα χρειαζόντουσαν και όσον αφορά τις καινούριες υποδομές και όσον αφορά τη συντήρηση παλιών. Και η τρίτη πρόκληση έχει να κάνει με τις συνδυασμένες μεταφορές. Ε, για σε εμπορικές μεταφορές τις οδικές έχουμε 45,8, για τις επιβατικές 73,7. Στις θαλάσσιες επίσης υπάρχει διαφορά 36,9 εμπορικές, 7,9 ε, επιβατικές. 80% όμως βλέπουμε ότι είναι οδικές τελικά. Και αυτή είναι επίσης μια πρόκληση η οποία έχει συμπεριληφθεί στις οικονομικές μας εκτιμήσεις. Ποια είναι τώρα η ευρωπαϊκή προσέγγιση. Τα διευρωπαϊκά δίκτυα άρχισαν ως προτεραιότητα των χωρών μελών σιγά σιγά από το 1996. Σήμερα έχουμε ένα οικονομικό εργαλείο αποτελεσματικό για πρώτη φορά γιατί έχουμε το τριπλό από ό,τι είχαμε παλιότερα. Βέβαια, εξαρτάται πώς το υπολογίζει κανείς. Είδαμε και τις προτεραιότητες και οι προτεραιότητες είναι σαφείς, τις βλέπετε στην επόμενη διαφάνεια και είναι για να δημιουργήσουμε ένα διευρωπαϊκό δίκτυο ε, καθορίσαμε εννέα βασικούς ε, διαδρόμους και πάνω σε αυτούς προετοιμάζουμε και τις επενδύσεις. Το μέσον που έχουμε στη διάθεσή μας το γνωρίζετε, να το. Έχουμε 26 δισεκατομμύρια στην αρχή για τη διευκόλυνση συνδέοντας την Ευρώπη και εδώ 11,3 που έρχονται από το Ταμείο Συνοχής. Οι προτεραιότητές μας στην προετοιμασία αυτή, στη χρηματοδότηση, είναι ότι είναι πιο περίπλοκο. Είναι οι συμφορήσεις, είναι οι διασυνοριακές διελεύσεις, είναι το διοξίδιο του άνθρακα, είναι οι συνδυασμένες μεταφορές οδικές, ε, σειροδρομικές, η διαλειτουργικότητα κλπ. Εδώ δηλαδή έχουμε καθορίσει διάφορα κριτήρια τα οποία δυσκολεύουν τον ευρωπαϊκό χώρο μεταφορών και που θα πρέπει να ξεπεραστούν για να πετύχουμε τον ευρωπαϊκό χώρο μεταφορών. Έχουμε δύο κανονισμούς, τον 1316 και τον 1315. Για τον 1316 βλέπετε εδώ ποια είναι η συγχρηματοδότηση. Βλέπετε τη συγχρηματοδότηση βάσει των ε, προτεραιοτήτων. Είναι η επόμενη διαφάνεια. Να, αυτή είναι. Αν δείτε λοιπόν τη συγχρηματοδότηση και πώς χρησιμοποιείται, θα δείτε ότι κατά μέσο όρο έχετε μια συγχρηματοδότηση 20 με 40% στις χώρες που δεν είναι συνοχής και μέχρι 85% στις χώρες συνοχής. Αυτό σημαίνει ότι η συγχρηματοδότηση αυτή που θα βγει από την διευκόλυνση συνδέοντα στην Ευρώπη είναι κάτι αναγκαίο για τη χρηματοδότηση ορισμένων έργων. Οι προτεραιότητες που έχουμε τώρα είναι οι διεπόμενες διαφάνειες καθορίζουν πολύ καλά τη σχέση ανάμεσα στα χρηματοδοτικά μέσα και τις προτεραιότητες που έχουμε καθορίσει για τις μεταφορές. Είναι στο πολιτές πρόγραμμα έτσι κι αλλιώς και είναι και στο ετήσιο πρόγραμμα. Προς το παρόν τα έργα τα οποία ήδη έχουν αρχίσει. Μέχρι το τέλος του 2014 έχουμε κάνει μια μελέτη διαδρόμων. Έχουμε και ένα σχέδιο εργασίας και επενδύσεων για τα πιο σημαντικά έργα. Και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή από τη δικιά της την πλευρά έχει κάνει έχει ήδη ζητήσει για ένα νέο έργο, κάτι το οποίο ολοκληρώθηκε τον Φεβρουάριο. Τώρα δηλαδή το μήνα που μας πέρασε. Μια έκκληση για προσφορές. Τώρα θα σας δείξω πόσα χρήματα βάλαμε και ποια είναι η απάντηση. Για το 2015 έχουμε εδώ την εκτίμηση αναδιάδρομο με τις προτεραιότητες της επενδύσεις μας και την αναθεώρηση που θα γίνει το 2017. Και εδώ έρχεται το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων, αυτή την επόμενη διαφάνεια. Με την διευκόλυνση συνδέοντας την Ευρώπη έχουμε το 8 δισεκατομμύρια. Και ο αντίκτυπος ποιος θα είναι, το βλέπετε εδώ. Το συνδέοντας την Ευρώπη με το νέο Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγών Επενδύσεων είναι 3,3 δις και για τις μεταφορές 2015 με 2018 έχουμε 2 δισεκατομμύρια, 2,7 δισεκατομμύρια με τα διάφορα άρθρα. Τα πιο σημαντικά άρθρα τα έχω εδώ. Είναι τα άρθρα που έχουν να κάνουν με τις συμφορήσεις, με τη χρηματοδότηση που προβλέπεται για τις εναλλακτικέ πηγές ενέργειας και το τρίτο είναι η διαλειτουργικότητα. Ποια είναι η σημερινή κατάσταση τώρα. Αν ξεκινήσουμε από την διευκόλυνση συνδέοντας την Ευρώπη, η κατάσταση είναι εξής. Αν βγάλουμε 2,7 δις για τα μέσα μεταφορές και η πρώτη πρόσκληση για την οποία σας μίλησα πριν που χρηματοδοτείται από τις χώρες μέλη με 8 δις και από το Ταμείο Συνοχής με 4 δις. Η πρόσκληση αυτή μέχρι τώρα, χωρίς να είναι οριστικό όμως, για 12 δις χρειάστηκαν 36 ε, δις, ζητήθηκαν δηλαδή για έργα. Είναι ενδιαφέρον ο προσανατολισμός αυτός αλλά μην το πάρετε οριστικό σαν νούμερο. Εκατό δις επενδύσεις σημαίνουν όλα αυτά. Η μόχλευση, θα έλεγα λοιπόν, είναι το 1 τρίτο. Αυτή είναι η δικιά μας διαπίστωση. Μπορώ να σας παρθιώσω και μια ανάλυση των έργων που προτάθηκαν στα πλαίσια του ταμείου που θα δημιουργηθεί. στα γρήγορα κάπως. Έγινε κάτω από τις σημερινέ συνθήκες που δεν είναι οι βέλτιστες, γιατί δεν έχουμε και αρκετό προσωπικό. Μεταφορές για 127 δις έργα έχουμε και για αυτά τα 127 δις τα μισά περίπου είναι για τις οδικές μεταφορές. Οι άλλες επενδύσεις είναι σιδηρόδρομοι, σύνδεση σιδηροδρόμων, όχι όμως υποδομές σιδηροδρόμων και αυτά μπορείτε να τα συγκρίνετε και με τις προτεραιότητές μας. Συγχρόνως αναλύσαμε και τις αδυναμίες που διαπιστώσαμε και εντοπίσαμε κατά το παρελθόν. Και εδώ έχετε τα συμπεράσματα μιας ομάδας εργασίας. Να τα τα συμπεράσματα. Γιατί υπάρχουν προβλήματα επενδύσεων στις μεταφορές. Το πρόβλημα είναι τεχνικό πώ θα υποβληθούν τεχνικά δηλαδή. Το δεύτερο είναι οι διευκρινήσει που χρειάζονται όσον αφορά τις κρατικές επιχορηγήσεις. Το τρίτο είναι οι στατιστικές όσον αφορά τις συμπράξεις δημοσίδιωτικού τομέα. Επειδή υπάρχει η συμπεριφορά των τραπεζών και υπάρχει και το πρόβλημα της αξιολόγησης. Ε, συμπερασματικά λοιπόν θα έλεγα ότι τα πρώτα μας συμπεράσματα είναι ότι διαπιστώνουμε πως η δημιουργία ενός βιώσιμου χώρου για τις μεταφορές χρειάζεται μια άμεση χρηματοδότηση 30%. Και η πρώτη πρόσκληση το αποδεικνύει αυτό. Αν δηλαδή μιλήσουμε για 12 δις και μας έρθουν αιτήσει για 36 δις που σημαίνει 100 δις επενδύσεις αυτό σημαίνει ότι βρίσκουμε το λογαριασμό έτσι. Έπειτα είπα ότι το πρόβλημα είναι η αξιολόγηση, η αξιολόγηση διαδρόμων. Συχνά υπάρχουν τα εθνικά συμφέροντα που εμπλέκονται σε κάθε έργο, χωρίς να δούνε το, τη σημασία που έχει ο διασυνοριακός παράγοντας. Τι μπορεί να βοηθήσει σε κάτι που γίνεται στην Αθήνα τον Βούργο, ας πούμε. Είναι αυτή η προσέγγιση διαδρόμων που είναι μια δύσκολη δουλειά. Έπειτα, ο κοινωνικός και οικονομικός αντίκτυπος. Οι επενδύσεις που γίνονται στους σιδηροδρόμους ή στις εσωτερικές πλωτές συγκοινωνίες. Κοινωνικά και οικονομικά ο αντίκτυπος είναι πιο μεγάλος από το καθαρά οικονομικό όφελος των επενδύσεων. Διοξίδιο του άνθρακα σας είπα ότι οι μεταφορές είναι μόνο στο μέσο που έχει αυξηθεί έχουν αυξηθεί οι εκπομπέ ε, διοξιδίου του άνθρακα. Δεύτερη κατηγορία συμπερισμάτων για τη συγχρηματοδότηση. Διαπιστώνουμε ότι ακόμα και στι χώρε συνοχή όπου υπάρχει 15-20% συγχρηματοδότηση, τελικά στο πλαίσιο της χρηματοδότησης αυτής υπάρχει πρόβλημα. Υπάρχει και το θέμα της εσωτερήκευσης του κόστους. Εδώ είναι μια συζήτηση που μπορεί να ανοίγει την πόρτα και στη σύμπραξη ιδιωτικού τομέα για κάποια έργα. Αλλά αυτή η εσωτερήκευση του κόστους ερμηνεύεται συγκεκριμένα σήμερα από το σύστημα διοδίων ε, και έχουμε τέτοια παραδείγματα. Αυτό σημαίνει επίσης ότι σε σχέδια τέτοιων συμπράξεων θα βρείτε περισσότερα έργα στον τομέα αυτόν από ό,τι αλλού όπου η επιστροφή δεν είναι ίδια, το κέρδος δηλαδή. Και το τελευταίο το οποίο διαπιστώνουμε είναι ότι θέλουμε με τους διαδρόμους αυτούς να θεραπεύσουμε κάποια οικονομία περιφερειακή, δηλαδή με το Ταμείο Συνοχής και με τα χρήματα της συνοχής για κάθε χώρα θέλουμε οι διαφορές που υπάρχουν στην οικονομική και κοινωνική εξέλιξη των περιφερειών να μειωθεί. Να μην λέμε δηλαδή ότι θα δανείζουμε μόνο ε, στους πλούσιους για να επενδύσουμε στις μεταφορές. Αυτή είναι προς το παρόν η προσέγγισή μας. Και σε αυτή τη βάση νομίζω ότι μπορούμε να κάνουμε μια καλή ανάλυση για την πρακτική δυνατότητα ε, χρησιμοποίησης του Ταμείου Αυτού Στρατηγικών Επενδύσεων. Οι προτάσεις είναι σίγουρα πολύ καλές. Πρέπει βέβαια να τις δούμε πιο λεπτομερώς και να τις δούμε και σαν πολιτική δράση και όχι μόνο σαν μια επενδυτική δράση και τελεία και παύλα. Και αυτό ακριβώς προσπαθούμε να κάνουμε και εμείς. Σας ευχαριστούμε κύριε Γκρός, ευχαριστούμε για αυτή την διαφωτιστικότατη ομιλία σας. Να δώσουμε τώρα το λόγο στους δύο συγκητές μας, κύριε Μπούλμαν, τρία λεπτά. Μετά, μετά μάλλον από τους ε, εισηγητές θα απαντήσουν οι δύο προσκεκλημένοι και μετά όσοι ξημών επιθυμείτε να λάβετε το λόγο έχετε τη δυνατότητα για 1,5 λεπτό. Μπούλμαν, ευχαριστώ. Ευχαριστώ βεβαίως τον κύριο Κέλλερ και τον κύριο Γκρό. Αρχίζω με εσά κύριε Κέλλερ. Κύριε Κέλλερ, η ιδέα που εκφράσατε ότι δηλαδή είναι δυνατόν ευφύς άνθρωποι να κάνουν υπορισμένες περιστάσεις να προχωρούν μάλλον σε λήψη ανόητων αποφάσεων μου φαίνεται τόσο πετυχημένη η παρατήρηση αυτή που θα τη θυμούμε. Το ερώτημα είναι τώρα πώς μπορούμε να αλλάξουμε τα πράγματα αυτά και κάτι είπατε σχετικά. Βέβαια υπάρχουν και ορισμένα προβλήματα στην μεταφορά του παραδείγματός σας σε αυτά που συζητούμε εμείς εδώ ως νομοθέτες. Μιλήσατε εσείς για σύστημα ανεξάρτητης λήψης αποφάσεων Βέβαια τόσο ανεξάρτητο το σύστημα δεν είναι εάν εξετάσουμε πώς λαμβάνονται οι αποφάσεις, ιδίως στην Επιτροπή, μάλλον στην ε, Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, η οποία στο παρελθόν έχει καταστήσει ιδιαίτερα σαφές ότι ενδιαφέρεται πρωτίστως για τον εαυτό της διότι εν τέλει έχει πει και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ότι δεν μπορεί το τριπλό α να είναι το μοναδικό κριτήριο για επιλογή. Το ΕΦΣΙ επίσης δεν είναι ανεξάρτητο ταμείο. Υπάρχει και μια συμφωνία μεταξύ αυτού που αναλαμβάνει την ευθύνη και που είναι ο Ευρωπαϊκός προπολογισμό και εκείνων που λαμβάνουν τις επενδυτικές αποφάσεις. Και εδώ είναι ασαφές το ποιος φοράει τα πανταλόνια, όπως λέμε. Δηλαδή το ποιος αποφασίζει το ότι πρέπει να υπάρξει ένας πολιτικός ηγετικός ρόλος για τον προσανατολισμό των επενδυτικών σχεδίων χωρίς αναπερίπτωση να ανακατεύεται αυτός που θα λαμβάνει τις αποφάσεις αυτές στην κάθε περίπτωση. Δεν το έχουμε ακόμα αυτό, ίσως αυτό να οφείλεται και στην νομοθετική μας διαδικασία. Για την ώρα όμως την ευθύνη φέρουν αυτοί οι οποίοι δεν αποφασίζουν. Τώρα για τον κύριο Γκρός. Πολύ ενδιαφέροντα τα όσα αναπτύξατε. Συγκεκριμένη ερώτηση. Από τα σχέδια που ε, συζητήσατε εσείς, ποια από αυτά μπορούν να χρηματοδοτηθούν από το ΕΦΣΥ. Το ΣΕΦ δεν θέλει από αυτά. Από τα συγκεκριμένα λοιπόν έργα που προτείνετε, ποια είναι δυνατόν να χρηματοδοτηθούν από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων. Λέτε ότι ορισμένα χρειάζονται μέχρι και 30% δημόσια χρηματοδότηση. Το ΕΦΣΥ δεν θα πρέπει να αρχίσει να συνηθίζει να σκέπτεται έτσι εάν θέλει να συναποφασίζει σε τέτοια πράγματα. Θα ήθελα να μάθω τη δική σας άποψη, αν έχετε ίσως και προτάσεις, πώς μπορεί να αντιμετωπίσει κανείς αυτή τη διάσταση. Ευχαριστώ. Φερνάντες. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ήθελα να σχολιάσω για τις δύο παρεμβάσεις που θα μας διευκολύνουν για να υποβάλουμε τις καλύτερες δυνατές προτάσεις και να βελτιώσουμε όσα προτείνονται για αυτό το Ταμείο Επενδύσεων. Η πρώτη μου ερώτηση για τους ομιλητές είναι η εξής. Το Ταμείο υποτίθεται ότι θα προσφέρει, θα αποφέρει μάλλον κέρδος. Είναι αδύνατο αυτή τη στιγμή να προβλέψουμε ότι κέρδο θα υπάρξει. Συμφωνώ με την ιδέα ότι το κέρδο αυτό θα πρέπει να προβλεφθεί, να, προ... να χρησιμοποιηθεί κιόλα και να αξιοποιηθεί για τα προγράμματα που θα έχουν πληγεί. Διότι πρέπει να πάρουμε την εγγύηση, όπως είπαμε, 16 δις ευρώ εκτιμάται ότι θα πρέπει να είναι, και να δημιουργήσουμε ένα ταμείο, 8 εγγύησης. Εκεί λογικό μου φαίνεται τα κέρδη να επιστρέψουν στον προπολογισμό για να ε, ενισχύσουν τις γραμμές που ενδεχομένως επλήγησαν αρχικά. Η δεύτερη μου ερώτηση έχει να κάνει με το Connecting Europe Facility. Ξέρουμε ότι ο στόχος του ταμείου αυτού βασίζεται στην αρχή της προσθετικότητας. Να συμπληρώσει δηλαδή όσα γίνονται αλλού δεν είναι υποκατάστατο. Απλώς θα επιτρέψει την κινητοποίηση των ιδιωτικών επενδύσεων. Εδώ υπάρχει μια σχετική σύγχυση. Κάποιοι θεωρούν σχεδόν αμαρτία τις ιδιωτικές επενδύσεις. Όχι, ιδιωτικέ επενδύσει για βιώσιμα έργα, για σταθερά έργα, για έργα που δημιουργούν θέσει απασχόληση και επιτρέπουν την ενίσχυση τη κοινωνική συνοχή, για προγράμματα που συνάδουν με την στρατηγική μα, την ε, στρατηγική τη Ευρώπη του 2020. Αυτέ οι ιδιωτικέ επενδύσει θα πρέπει να ε, ενδυναμωθούν. Συγκεκριμένη ερώτηση όμω, πώ μπορεί να συμβαστεί το ΕΦΣΙ με την αρχή της προστατικότητας και συγκεκριμένα με τις επενδύσεις που γίνονται ούτως ή άλλως μεταξύ του ε, Connecting Europe Facility και των διευρωπαϊκών δικτύων μεταφοράς. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Φερνάντες. Καλό τον κύριο Κέλλη να απαντήσει στους δύο συγκεκριτές μας. Δύο λεπτά παρακαλώ. Ευχαριστώ, Ευχαριστώ πολύ. Να αρχίσω απαντώντας στον κύριο Μπούλμαν. Συγκεκριμένη σύσταση θα μπορούσε να είναι η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων να χρηματοδοτήσει συγκεκριμένες πλατφόρμες. Πλατφόρμες οι οποίες μετά θα χρηματοδοτήσουν την επανευθυγράμμιση κάποιων κινήτρων. Αυτό είναι κάτι διαφορετικό από το να συμπληρωθούν ιδιωτικές επενδύσεις. Κανείς από τους ιδιώτες χρηματοδότες δεν, ιδιώτες επενδυτές δεν χρειάζονται δημόσια χρήματα. Τα χρήματα του δημοσίου, δανεισμός από το δημόσιο δηλαδή, κοστίζει πολύ, έχει πολύ ψηλό κόστος και δεν το χρειάζεται κανείς. Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων μπορεί να χρηματοδοτήσει πλατφόρμες, το KENAP μπορεί να είναι μια τέτοια πλατφόρμα, υπάρχουν όμως και, πολλοί άλλες, και πολλές άλλες που μετά αυτές θα επενδύουν σε μια ευθυγράμμιση των κινήτρων για να αλλάξουν μη αποδοτικές βιομηχανικές δομές που έχουμε σχέση για παράδειγμα στον ε, κλάδο των ιδιατρικών βιομηχανικών στην Ευρώπη καθώς και για να αντιμετωπιστούν ελλείμματα της εμπλοκής της κοινωνίας των πολιτών που πάλι οδηγεί με τη σειρά του σε ε, βαχνορισμένα κενά των επενδύσεων αυτών. Για παράδειγμα, για τα εμβόλια. Υπάρχει πραγματική ευκαιρία και δεν χρειάζεται διαφορετική διακυβέρνηση. Απρός πρέπει να γίνουν ε, οι σωστές αποφάσεις για τις επιχειρήσεις μέσω της πλατφόρμας των επενδύσεων και με εγγυήσει που θα καλύπτονται. Αυτό με φέρνει στο δεύτερο σημείο, ότι όπως είπατε κι εσείς, βεβαίως ε, έχει νόημα να αποφέρουμε κέρδος ο κάθε επαγγελματία και ο κάθε επενδυτή θέλει να βγάλει κέρδο. Απλώ το θέμα είναι ποιε είναι οι δυνατότητε διαχείριση που έχουμε κι εμεί. Και αυτά τα κέρδη σε κάθε περίπτωση πρέπει να αξιοποιηθούν για να αλλάξει η διάρθρωση του Ταμείου. Δεν είναι τόσο περίπλοκο και θα πρέπει, δεν θα χρειαστεί να πεινώσουμε ξανά τον τροχό. Στην πραγματική αγορά τα εργαλεία υπάρχουν. Αυτό που χρειαζόμαστε είναι διαφορετική διάρθρωση. Δηλαδή το ΕΦΣΙ και η ΕΤΕ με ένα λογικό τρόπο ε, να επικεντρωθούν σε αυτό που μπορούν να κάνουν ε, πραγματικά. Ε, ο Εμιλητής μας είπε μια στα γερμανικά που δεν μπορούμε να μεταφράσουμε. Κύριε Γκρός, θα μιλήσω στα γερμανικά. Η ερώτησή σας για το ποια ε, έργα μπορούν να χρηματοδοθούν απευθείας να δώσω μια απάντηση με διαφορετικές ε, αποχρώσεις, δηλαδή δεν έχει τόσο πολύ σχέση με το τι μόχλευση θέλουμε να πετύχουμε η επιλογή. Χρειαζόμαστε 80% επενδύσεις στους σιδηροδρόμους. Υπάρχει πραγματικό έλλειμμα στους σιδηροδρόμους σε όλες τις χώρες και οι σχετικές επενδύσεις λείπουν. Εάν υπάρξουν, Θα υπάρξει κέρδος, αλλά όχι εγγυημένο. Να σας δώσω ένα παράδειγμα των ε, επενδύσεων με τις εναλλακτικές μορφές ενέργειας. Για παράδειγμα, για λιμάνια κλπ. Όπου λείπει η υποδομή αυτή και να επιτρέψει η υποδομή αυτή και τη μετάβαση σε εναλλακτικές ενέργειες. Μπορεί να μείνει κανείς εδώ ότι η βιομηχανία και αν συμμετάσχουν και ορισμένοι τομείς μπορεί να αναζητήσει τις εταιρικές αυτές σχέσεις. Όχι λοιπόν στις μεγάλες επενδύσεις, αλλά στις μικρές αυτές επενδύσεις ναι, είναι δυνατό αυτό. Τέλος, τι είδους μορφή κινητικότητας θέλω εγώ και αν υπάρχουν τα σχετικά εργαλεία για να διεξαχθεί η πολιτική αυτή ή αν υπάρχουν τα εργαλεία για να υποστηριχθούν επενδύσεις χωρίς, κάποια, χωρίς να δοθεί άνωθεν κάποια κατεύθυνση. Έχει το λόγο εσείς τώρα κύριοι συνάδελφοι όσοι επιθυμείτε να εκφράσετε άποψη. Βάλει. Ευχαριστώ. Μια συντομότατη ερώτηση. Για το συντονιστή των διευρωπαϊκών δικτύων. Δεδομένου ότι το πρόγραμμα Juncker θα πάρει κονδύλια από προγράμματα που χρηματοδοτούν τον Ευρωπαϊκό Προπολογισμό για να πάνε τα κονδύλια αυτά στις εγγύησεις. 700 εκατομμύρια θα αφαιρεθούν από το Connecting Europe Facility. Για λόγους ανεξάρτητου συμβουλίου ή ε, χαμηλής ε, απόδοσης των επενδύσεων στις υποδομές ή τη χαμηλή διάθεση να υπάρξουν επενδύσεις σε αυτό το τομέα. Το εύση... ποιες, ε, μάλλον στην αθαίρεση των κονδύλιων, ποια έργα θα παραμείνουν ε, στο περιθώριο και δεν θα χρηματοδοτηθούν. Ο κύριος Ρικέ από την Επιτροπή Μεταφορών, πρόεδρε, θα εκφραστώ ως ε, πολιτικός και ερετός που είμαι και όχι ως ειδικός εμπειρογνώμων που δεν είμαι. Μία ερώτηση προς τον κύριο Κρός. Μας, ε, νομίζω ότι εδώ έγινε μια παρανόηση, διότι δεν νομίζω ότι μπορούμε να περάσουμε από ένα δημοσιονομικό εργαλείο σε ένα άλλο με τις ίδιες πολιτικές και να τις κάνουμε αποτελεσματικότερες. Αυτό που θα κάνουμε είναι να, πά, να αλλάξουμε ε, μέσο και εργαλείο, μηχανισμό, για να πάμε από ένα είδος πολιτική σε ένα άλλο. Αυτό νομίζω προσπάθησε να μας εξηγήσει ο κ. Γκρός. Δηλαδή τα προγράμματα του Horizon 2020 και του Connecting Europe Facility είναι προγράμματα πολιτικής, για τα οποία όμω δεν υπάρχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον από του ιδιώτες επενδυτές καταλαβαίνουμε την ανάγκη να περάσουμε σε ψηλότερα επίπεδα ε, κρατική χρηματοδότησης. Ε, έτσι, αν δεν υπάρξει αυτό, δεν θα υλοποιηθούν τα προγράμματα. Στο Κοινοβούλιο τα συζητούσαμε επί χρόνια τα προγράμματα αυτό για να λάβουν τον ανάλογο χαρακτηρισμό, για να πάρουν την ευρωπαϊκή προστιθμένη αξία που τους αξίζει, για να συμφωνούν με τις πολιτικές περιβάλλοντος, τις κοινωνικές, τις οικονομικές αυτό που θα βγάλουμε από το Horizon 2020 και, θα το βάλ, και από το Connecting Group Facility για να το βάλουμε στο ταμείο, είναι κάτι που παίρνουμε από μια πολιτική για να το βάλουμε σε μια άλλη. Δεν κάνουμε καθόλου την ίδια πολιτική μεταφορών ή έρευνα, όπω πολύ σωστά εξηγήθηκε από του ομιλητέ με το EFSI ή με το Connecting Euro Facility ή με το Horizon 2020. Αυτή ήταν η πρώτη μου παρατήρηση και η δεύτερη ήταν ότι το βρίσκω πραγματικά περίεργο στις δημοσιονομικές αρχές. Εδώ η δημοσιονομική αρχή εκπροσωπείται πολύ καλά από την Επιτροπή Προπολογισμών και την Επιτροπή και του συναδέλφους. Εδώ λοιπόν τους ε, επιβάλλουμε ε, μια διάλυση των δημοσιονομικών πολιτικών που προβλέπετε. Μου φαίνεται πραγματικά ε, απίστευτο. Του λέμε θα βάλουμε χρήματα σε ένα ντουλάπι από τα οποία η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα υποφεληθεί με ένα συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα και ε, άσχετα με τη γνώμη τη δημοσιονομική αρχή. Πρώτον δηλαδή αλλάζουμε πολιτική και δεύτερον αναλαμβάνονται δημοσιονομικές αρμοδιότητες τελείω αυθαίρετε δημιουργώντα ένα ταμείο τραπεζικό στην ουσία. Εδώ ήθελα να δώσω να κάνω μια ερώτηση στον κύριο Γκρός που υπήρξε και βουλευτής και ξέρει πολύ καλά το σύνολο των θεμάτων αυτών. Θα εφαρμοστεί η ίδια πολιτική μεταφορών και έρευνας με τα εργαλεία που όλοι μαζί καθορίσαμε με δουλειά εδώ και μια τετραετία Όπω για τα δημοσιονομικά εργαλεία που είχαμε τώρα, θα γίνουν τα ίδια για το ταμείο που συζητάμε. Ευχαριστούμε, κύριο Σκάρα. Κύριε Πρόεδρε, μου άρεσαν τα πρακτικά παραδείγματα που έδωσαν. Γιατί χρειαζόμαστε για κάποια benchmark. Μου άρεσε επίσης που άκουσα από τον κύριο Κέλλερ και που ξεφύγαμε λίγο από αυτή την καθημερινή συζήτηση για την οδηγία και τον κανονισμό, διότι το κέριο ερώτημα είναι τι είδου Ευρώπη θέλουμε εν τέλει. Σε ποιου τομεί θέλουμε να γίνουμε ηγέτες της παγκόσμιας αγοράς. Πού έχουμε τι μεγαλύτερες ελλείψεις. Αν τα βρούμε αυτά θα ξέρουμε σε ποιους τομείς θέλουμε να επενδύσουμε. Βεβαίω και χρειάζονται εδώ κάποια ειδικά, ειδικότερα στοιχεία. Το γεγονός όμως ότι θα προσελκύσουμε το ιδιωτικό κεφάλαιο μόνον εάν η απέτηση για ανεξάρτητε αποφάσεις, η απέτηση για global player, η απέτηση για ένα συνολικό όραμα, αν δεν υπάρχουν αυτά, τότε δεν θα προσέλθουν οι ιδιώτες επενδυτές. Θα ήθελα να μάθω τον κύριο Κέλλερ. Πού βλέπετε την διασύνδεση μεταξύ του δικού σας ιδιωτικού του δικού σας ταμείου και του EFSI. Και υπάρχει κάποια δυνατότητα συνεργασία των δικών σας προγραμμάτων με τον ΕΦΣΙ. Και κατάλαβα καλά ότι βλέπετε μια διασύνδεση μεταξύ ημών και του κ. Γκρός. Έχετε μια πλατφόρμα μεταφορών. Έχετε μια πλατφόρμα για να εργα... για ενέργειες όπου να επι τρέψει έτσι την οικοδόμηση μιας γέφυρας μεταξύ των δυο σας. Και η Διευθυντική Επιτροπή θα πρέπει να συναπαρτίζεται από πρόσωπα που είναι ανεξάρτητες προσωπικότητες και δίνουν έτσι το μήνυμα στους ιδιώτες επενδυτές ανεξάρτητα από το που εντάσσονται πολιτικά. Ευχαριστώ. Η κυρία Αιάλα Σέντερ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα, στις συζητήσεις που κάναμε αυτές τις μέρες για το EFSI, ακούγεται κάτι που μένα με ανησυχεί. Ότι από την πρόταση Κέλλερ, που μου φαίνεται βέβαια ελκυστική, ένα από τα κριτήρια είναι η ανάγκη αλλαγών στην τρέχουσα νομοθεσία. Διάβασα λίγο για την πλατφόρμα Κενούπ και φαίνεται ότι πρόκειται για αλλαγές στην νομοθεσία. Αυτό, τι να σας πω εμένα, με ανησυχεί. Γιατί το νομοθετικό πλαίσιο είναι αυτό που είναι. Μπορούμε να κάνουμε κάποιες προσαρμογές, αλλά τέτοιες αλλαγές θέλω να ρωτήσω πώς ακριβώς θα έχουν για να μην συνεχίζονται τα λάθη. Στον κύριο Κρός θέλω να πω ότι πάντα στα πλαίσια αυτά του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων τι γίνεται με το Solvency 2, το Βασιλεία 3, δηλαδή υπάρχει ανάγκη να αλλάξει κάπως η βάση εδώ στο Κοινοβούλιο. Και το λέω και στους συναδέρφους για να γνωρίζουμε για τι πράγμα μιλάμε. Γιατί μας δίνουν μερικές φορές χρήματα με το ένα χέρι, αλλά από την άλλη μεριά μας εμποδίζουν να νομιθοποιούμε. Τώρα μας μιλήσατε πολύ για την δυνατότητα χρηματοδότησης απ' έξω. Κίνα, μπορεί να είναι και Ρωσία, δεν ξέρω. Εσείς πώς το βλέπετε αυτό το θέμα της χρηματοδότησης απ' έξω. Και στον κύριο Γρός για τη χρηματοδότηση του Πακού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων. Ο κύριο Μάιστατ μα είπε ότι υπάρχει κίνδυνο γεωγραφική συγκέντρωση και κίνδυνο τα κίνητρα να είναι αναχώρα για αυτές που είναι κάτω από 3% μία χώρα ή τέλο πάντων περισσότερες. Θέλω να ξέρω, υπάρχουν τέτοια κριτήρια που γνωρίζετε εσείς για τα κίνητρα. Και τέλος όσον αφορά τις Επιτροπές Εμπειρογνωμόνων. Ποιοι θα είναι αυτοί και θα είναι γιατί αποφάσεις που όπως είπε και ο κύριος Μπούλμαν δεν θα στέκουν. Γιατί την τελική, η τελική απόφαση φοβούμαστε ότι θα καταστρέφει τις αρχικές προτάσεις τελικά. Πρόεδρος, έχουμε τους εισηγητές μεταξύ μας της Επιτροπής Περιφερειών και της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής. Τον κύριο Γκέβετ, αν θέλει να παρέμβει. Α, έφυγε στο μεταξύ. Ο κύριος Σμιθ, που είναι εισηγητής από την ΟΚΕ, είναι εδώ. Όχι. Καλά, τι να κάνουμε. Του χαιρετίζω, αν και έφυγαν. Ήταν όμως εδώ ένα μεγάλο κομμάτι. Δεν έχει ζητήσει κανένας άλλος το λόγο. Σωστά. Συνεπώς, θα δώσω το λόγο στους προσκεκλημένους μας, στους ομιλητές μας δηλαδή, για να απαντήσουν. Πρώτα, ο κύριος Κέλλερ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Επιτρέψτε μου να δομήσω κάπως την απάντησή μου. Τι προσπαθούμε να προτείνουμε ότι το Κοινοβούλιο πρέπει να δει την νομοθεσία για επενδύσεις προς την πλατφόρμα επιχειρήσεων. Δεύτερον, για την δικιά σας την ερώτηση. Η πλατφόρμα αυτή επενδύει βάσει κινήτρων και βάσει εξυγχρονισμού της νομοθεσίας. Αυτό βέβαια έχει να κάνει όταν μιλάμε για την τεχνολογία εχμής και δουλεύουμε με εργαλεία και με μέσα που τα έχουμε κληρονομήσει από τις δεκαετίες του 50 και του 60. Πώς είναι δυνατόν λοιπόν να ρυθμίσουμε ε, πράγματα που έχουν να κάνουν με πιο πρόσφατη τεχνολογία για παράδειγμα για εμβόλια τα οποία είναι σημερινά. Πώς είναι δυνατόν να προσαρμοστούμε με τέτοια παλιά εργαλεία. Θα μπορούσαμε να είχαμε διάφορα εμβόλια κατά του καρκίνου που σίγουρα περιπλέκουν πολύ περισσότερο την κατάσταση. Η επιστήμη δηλαδή πολλές φορές βρίσκεται πολύ πιο μπροστά από τις νομοθετικές ρυθμίσεις. Υπάρχουν 69 ρυθμιστές ε, για τα εμβόλια, για παράδειγμα, στην Ευρώπη, στην Αμερική ένας μόνο. Οπότε, απλές προσαρμογές μπορούν να έχουν τεράστιο ωφέλη. Δεύτερον, αν δούμε το Ευρωπαϊκό Σύστημα Καινοτομίας, αυτό που διαπιστώνουμε είναι ότι δεν υπάρχει αρκετή χρηματοδότηση ούτε προσαρμογές. Ας δούμε το Horizon 2020 ή άλλα αντίστοιχα προγράμματα. Πριν να υπάρξει μια ευκαιρία για ιδιωτικές επιχειρήσεις, υπάρχει ένα τεράστιο κενό στην Ευρώπη, πολύ περισσότερο από ό,τι οπουδήποτε αλλού στον κόσμο. Εδώ το Ταμείο λοιπόν μπορεί να παίξει ουσιαστικό ρόλο έστω και δευτερευόντως, ενθαρρύνοντας διάφορα μέσα και εργαλεία, προκειμένου να υπάρξουν επενδύσεις. Τέταρτον, όταν μιλάμε για σύμπραξη δημοσίου τομέα, πρέπει να ξέρουμε ότι τέτοιες επενδύσεις δεν θα λειτουργήσουν. Αυτό που μπορείτε να κάνετε είναι ή να δουλέψετε με συμπληρωματικές με συμπληρωματικά μέτρα, βιομηχανίες με επενδύσεις εντατικές, πρέπει να ξέρετε ότι οι εμπορικές επενδύσεις προωθούνται έτσι. Οι ανταγωνιστικές επενδύσεις προωθούνται. Κύριε Κάρα και για τη δικιά σας την ερώτηση, αυτό που προτείνουμε σήμερα δεν είναι απαραίτητα κάτι για την υγεία. Είναι ένα απλό παράδειγμα η υγεία. Προτείνουμε ένα σύστημα που μπορεί να προσαρμοστεί και σε άλλους κλάδους. Εφόσον βασίζονται στην έρευνα πολύ και έχουν ε, τεράστιες δυνατότητες ανάπτυξης και δεν πρόκειται για επενδύσεις παραδοσιακά δημόσιου τομέα. Και ναι, απάντηση στη δεύτερη ερώτησή σας, μπορούμε να κάνουμε πολύ περισσότερα με εγγύηση είτε από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων είτε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Κέλλερο. Κύριος Γκρός τώρα. Συνοψίζοντας, για να απαντήσω στην ερώτηση αν το EFSI μπορεί να κάνει την ίδια πολιτική με την διευκόνηση συνδέοντα στην Ευρώπη, μπορώ να πω ότι αν το EFSI προσαρμόσει τα κριτήρια, τις προτεραιότητες για τα διευρωπαϊκά δίκτυα, τότε μπορεί ναι. Εάν στο άρθρο 5 δεν θεσπιστούν τα κριτήρια αυτά, θα υπάρχουν άλλες προτεραιότητες, όχι όμως οι προτεραιότητες που έχουμε στο επίπεδο της διευκόλυνσης συνδέοντα την Ευρώπη. Είναι σαφές αυτό. Υπάρχει μια ζήτηση επενδύσεων, επανέρχομαι σε αυτό που είπαμε σε ορισμένες χώρες μέλη, για παράδειγμα Γερμανία. Και αν πάρω μονάχα τους δρόμους, στη Γερμανία. Σύμφωνα με μια ανάλυση του 2012 υπάρχει μια ανάγκη επενδύσεων της τάξης των 7 δισεκατομμυρίων ευρώ. Δεν, υπάρχουν, δεν υπάρχει έλλειψη λοιπόν της ζήτησης αυτής, είναι όμως προς προσανατολισμοί. Είναι σαφές αυτό και νομίζω ότι απαντώ έτσι στις δύο πρώτες ερωτήσεις. Σε ό,τι αφορά την γεωγραφική συγκέντρωση, νομίζω ότι είναι τα κριτήρια της χρέωσης που ισχύουν μέχρι τώρα. Αυτά τα οποία θα υπαγορεύσουν την συγκέντρωση. Ακόμα και στις χώρες όπου συγχρηματοδότηση του 15% του 20% ζητείται, ακόμα και εκεί μπορεί να προκληθούν προβλήματα. Εάν μπούμε λοιπόν σε αυτή την οπτική των, των ακριβών δημοσιονομικών κανόνων, είναι σαφές ότι η παρούσα πρόταση θα συμβάλλει να συγκεντρωθούν οι επενδύσεις σε ορισμένες χώρες μέλη και να αφήσουν απ' έξω άλλες. Για το περίφημο global player, θα ξανάρθω στο παράδειγμα αυτό, έχουμε χάσει από εδώ και πολύ καιρό ένα πολύ ξεκάθαρο, δηλαδή ότι ο σιδηρόδρομος μπορούσε να γίνει global player και μια κατεξοχήν ευρωπαϊκή επένδυση. Και τι γίνεται τώρα? Από τον τομέα που εργάζομαι, αν πάρετε το τρένο στο Αμβούργο για να πάτε στην Αθήνα, θα πρέπει να αλλάξετε τέσσερις φορές την ε, μηχανή έλξεως, εφτά φορές το βολτάζ. Αν πάρω το ε, φορτηγό όμως, θα χρειαστεί μόνο να σταματώ στα βενζινάδικα για να φορτώνω ε, πετρέλαιο. Αν λοιπόν αύριο θέλουμε να γίνουμε global player, θα χρειαστούμε ένα ευρωπαϊκό τρένο μεγάλης ταχύτητας. Έχουμε το ITS στη Γερμανία, να το έχουμε σε όλη την Ευρώπη. Άρα πρέπει να δώσουμε σήμερα τι δυνατότητε στη βιομηχανία που και αυτή μετράει μερικές χιλιάδες θέσει εργασία, Βέβαια υπάρχει ο κινέζικος και ο ιαπωνέζικος ανταγωνισμός να μπορέσει η βιομηχανία να επενδύσει για να φτιάξει αύριο το Airbus που θα κινείται πάνω στις ράγες. Είναι μια επένδυση με τεράστια προστιθέμενη αξία για την Ευρώπη και για τη βιομηχανία και για την κινητικότητα. Αν λοιπόν θέλετε να ψάξετε να βρείτε ένα έργο που να αξίζει την επένδυση, να το. Μα μένουν τέσσερα λεπτά. Θα, θα θέσω κάποιες ερωτήσει. Διότι για ορισμένα έργα βλέπουμε ότι η κερδοφορία τους θα προκύψει αν υπάρξει σταθερότητα στο ρυθμιστικό πλαίσιο. Αναφέρατε του σιδηροδρόμου. Εάν δεν το σχεδιάσουμε ξανά το ρυθμιστικό πλαίσιο, οι επενδυτέ μπορεί τουλάχιστον να έχουν επιφυλάξει. Διότι χωρί ε, το κατάλληλο ε, ρυθμιστικό πλαίσιο δεν θα έχουμε κατά την κερδοφορία και για τα φάρμακα που αναφέρατε εσεί ε, κύριε Κέλλερ, εάν οι δημόσιες αρχές δεν χρηματοδοτήσουν για να στηρίξουν τις χώρες που χρειάζονται αυτά τα φάρμακα, οι επενδυτές θα είναι τουλάχιστον επιφυλακτικοί. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρξει συντονισμός μεταξύ των πολιτικών αρχών και της ρυθμιστικής κατεύθυνσης που θα λάβουμε. Να θυμίσω το τι έγινε με τα φωτοβολταϊκά πάνελ ε, τελευταίως. Εάν δεν υπάρχει κάποια προστασία κατά του dumping των εξαγωγών, αρκετοί επενδυτές δεν θα αναλάβουν δεσμεύσεις. συμφωνώ απολύτω, αλλά για τι μεταφορέ αυτό που μπορώ να πω είναι ότι υπάρχουν ήδη κείμενα επιτάπητο και μπορεί να προκύψει το ρυθμιστικό πλαίσιο που να είναι πολύ περισσότερο αξιόπιστο. Να θυμίσω το τέταρτο πακέτο, την τέταρτη δέσμη μέτρων για του σιδηροδρόμου. Υπάρχει και ένα τεχνικό πυλώνα, ο οποίο ακριβώ ζητάει αυτό που σα είπα προηγουμένω, τη διαλογικότητα των τεχνικών συστημάτων μεταξύ των χωρών. Οι, οι χώρε μέλη λοιπόν έχουν το δικαίωμα. Δεν είναι η συζήτηση εύκολη γιατί ο καθένα θέλει να διατηρήσει τι εθνικέ του προαιρέσει. Αλλά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Κοινοβούλιο ε, έχουμε κάνει το καθήκον μα προετοιμασία του ρυθμιστικού πλαισίου. Λέω για τι μεταφορέ βέβαια. Ε, η αποτελεσματικότητα των χρηματοδοτικών εργαλείων αλλά και της, ε, των εκματικού πλησίου θα εξαρτηθεί από τα κάτι μέλη και από την καλή τους διάθεση. Αυτό νομίζω ότι μπορεί να είναι μια γενική έκκληση όχι μόνο για τις ε, μεταφορές που θα μπορούσαμε να απευθύνουμε και προς το Συμβούλιο. Και ίσως είναι και ένας τρόπος να αποπερατωθεί η εσωτερική αγορά μειώνοντας τον ρυθμό των ρυθμιστών όπως και για τις τηλεπικοινωνίες. Ε, κύριε Κέλλερ, παρακαλώ. Ευχαριστώ. Συμμερίζομαι τα προβλήματα των σιδηροδρόμων, γιατί εκεί βουλάει η σύζυγό μου, αλλά στους γερμανικούς σιδηροδρόμους. Όμως, ε, εδώ η λογική μα θα πρέπει να είναι η εξή. Να δημιουργήσουμε ευκαιρίε για τις νέες εταιρείε με καινοτομία και νέες ε, προσφορές μέσω των ε, πρωτοπόρων λύσεων, με υποψηφίου, για μεγάλε μορφέ συνεργασία. Σε πολλές ε, περιπτώσεις επιχειρήσεων ε, που είναι, θα μπορούσαν να αναλάβουν δράση σε αυτούς τους τομείς, η Ευρώπη έχει πολύ χαμηλό ποσοστό νεοφιών εταιριών. Εδώ λοιπόν η βασική μας αρμοδιότητα είναι να δημιουργήσουμε τέτοια ρυθμιστικά συστήματα που να στηρίζουν τις χώρες όπου υπάρχει καινοτόμο πλαίσιο εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης και να μεγαλώσουν οι νεοειδρυφείς επιχειρήσεις σε τομείς που ενδιαφέρουν ιδιαίτερα στην Ευρώπη ως προς την οικονομική ανάπτυξη. Πρέπει να γίνει μια άκοπη προσπάθεια για να δούμε ποιες επιχειρήσεις είναι αυτές που χρειάζονται τη στήριξή μας και τι συγκεκριμένα πακέτα θα απευθύνουμε προς την καθεμιά. Υπάρχουν πολλές δυνατότητες και σε άλλους τομείς εκτός από τους Ευχαριστώ. Φτάνουμε στο τέλος για την ε, διαλογικότητα ιδίω των σιδηροδρόμων. Νομίζω καλά ήταν ε, αυτό το τελευταίο σημείο που θίξαμε. Ε, τώρα, η επόμενη συνεδρίασή μα είναι στο Στρασβούργο, 5η-12 Μαρτίου, από τι 8 έω τι 10. Και θα είναι μια μεγάλη στιγμή, διότι στι 12 Μαρτίου θα μα παρουσιαστεί το σχέδιο έκθεση. Κύριοι συγητές, Έχετε την εμπιστοσύνη μας και ελπίζω ότι η σημερινή ακρόαση θα είναι για σας ε, κάτι που θα σας εξυπηρετήσει στην ε, δουλειά σας. Ρομπέρτο. Νομίζω ήταν εντατική ημέρα, οπότε μπορούμε να κηρύξουμε τη λήξη της συνεδρίασης. Και βεβαίω, κοιτάζοντα και περιμένοντα από του εισηγητέ, τους και την υποβολή τη εκθεσή του την επόμενη εβδομάδα στο Στρασβούργο. Σα ευχαριστώ. Καλό σα βράδυ.